Ο Πρόεδρος, κυρίες και κύριοι, πρώτα-πρώτα συμπαθάτε με, γιατί αρχίζουμε καθυστέρηση, γιατί τελείωσε ο πρώτος ε, όσον αφορά ε, τις τηλεπικοινωνίες πριν από λίγο. Η κυρία Κασίγια Βέρα ήταν ε, είχε τον πρώτο λόγο τέλο πάντων εκεί, η κυρία Πατρίτσια Τρόια, η Τόια ήταν εκεί και πήρε Επομένω, αυτέ οι δύο κυρίες οι οποίε μα εκπροσωπούσαν βέβαια, έχουμε και άλλους ε, συναδέλφους, του και ηγητέ. Οπότε μάλλον πρόκειται περί επιτυχίας. Δεν ξέρω αν η Πατρίτσια ε, πρεσβεύει τα ίδια. Α, βλέπω, γνέφηκα τα φατικά. Ωραία, ωραία. Πάντως ε, έχουν μπροστά μας πολλή δουλειά. Ιδίω όσον αφορά τα θέματα του βρυζονικού φάσματος, είναι κάτι το οποίο ακόμα δεν κρίθηκε στο Συμβούλιο και αυτό θα είναι για μας ένα μεγάλο πρόβλημα. Αλλά ίσως έχουμε και άλλα θέματα τα οποία θα πρέπει να επιληθούν. Δεν ξέρω τι σημαίνουν όλα αυτά για το μέλλον και τι μας επιφυλάει στο μέλλον. Δεν ξέρω, ε, ένα χρόνο θα περιμένουμε την ε, ε, κοινή θέση ένα χρόνο την περιμέναμε, θυμάστε, να δούμε τι θα γίνει τέλο πάντων. Αλλά οπωσδήποτε να διατηρούμε την αισιοδοξία μα. Συνάδελφοι, η μέρη σε διάταξη. Θέλει κανεί κάτι να αλλάξει, όχι από ό,τι φαίνεται. Και για τα διάφορα. Α, αυτό είναι το τελευταίο. Απλώ γίνω του Πρόεδρου θέλω να σα πω ότι βάσανε οι συντονιστέ να ματιώσουν την συνεδρίαση της Δευτέρας 13. Α, μισό λεπτό ήταν ο κύριος ε, Σεύκοβιτς. Ε, καλώς ορίσατε. Πρόεδρε, μισό λεπτό γιατί πρέπει να δούμε κάποια πρακτικά ζητήματα. Ε, Δύο-τρία λεπτά και όχι παραπάνω. Οπότε, 13 Τετάρτου. 13 Τετάρτου, η απογευματινή συνεδρία θα ματιωθεί επίσης όσον αφορά αυτήν την πρωτοβουλία που θα τη συζητούσαμε αυτήν την ε, ημερομηνία, στις 13 Απριλίου δηλαδή, θα την συζητήσουμε την Δευτέρα 20 Απριλίου. Απόγευμα, 3 με 6.30. Θα γίνει η συνεδρίαση όπως προβόταν για την 3η 14 Απριλίου. Έχετε λάβει και ένα σχετικό έγγραφο. Οι δε την Τρίτη 9 με 10 που με σε τακτική συνεδρίαση θα γίνει αύριο 24 Μαρτίου στις 10 η ώρα με ψηφοφορίες τι οποίε θα διεξαγάγουμε αύριο επομένως πολύ σημαντική ημέρα και αρχίζουμε 10 η ώρα λέει ο κάτι άλλο τώρα σημαντικό σας μενημίζω ότι συγκροτήθηκε ομάδα εργασία για την ψηφιακή Ευρωπαϊκή Ένωση την ε, Πέμπτη. Και σας κοινοποιήθηκε αυτό το σχετικό έγγραφο. Επίσης έχω να σας πω ότι η συγκρότηση σε σώμα θα γίνει την Πέμπτη, αυτή τη βδομάδα. Σε τρεις μέρες. Στις 26 Μαρτίου δηλαδή, 11 με 12 και 30. Η συγκρότηση σε σώμα αυτής της ομάδας εργασίας. Επίσης, θα χωριστεί στα δύο η συνεδρίαση. Πρώτα πρώτα η συγκρότησε σώμα και θα συζητήσουμε το, το πώς οι εργασίες και κατά δεύτερο λόγο στη συνέχεια θα συζητήσουμε με τον Ρόμπερτ Μάντελιν της ε, αρμόδιας γενικής διεύθυνσης τον οποίο τον έχουμε προσκεκλημένο, αλλά θέλω και εσείς όλα τα μέλη της Επιτροπής μας να έρθετε σε αυτή την συνεδρίαση και ενεργά να συμμετάσχετε σε αυτή την συζήτηση για τα ψηφιακά. Για τη ψηφιακή οικονομία, ψηφιακή ένωση συναλλαγές τηλεπικοινωνίας, Όλα αυτά θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και θα τα συζητήσουμε κατά την συνεδρίαση. Αυτά. Τώρα στο τρίτο σημείο έχουμε την έγκριση των πρακτικών. Έχετε λάβει τα πρακτικά. 21η-22η Ιανουαρίου και 26η Ιανουαρίου του 2015. Αν δεν υπάρχει κάποια ένσταση, τότε θεωρώ ότι εγκρίνονται τα πρακτικά. Όπως θυμάστε, κάναμε μια άτυπη συνεδρίαση στο Στρασβούργο. Είχαν συμμετάσχει οι επίτροποι και όμως δεν προβλέπονται πρακτικά για την άτυπη συνεδρίαση, την έκτακτη συνεδρίαση. Και πάμε τώρα στο τέταρτο σημείο. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση της ενεργειακής στρατηγικής ένωσης, ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, αρμόδιο για την Ενεργειακή Ένωση, τον κύριο Μάρος Σεύτσοβης. Σας ξαναβλέπουμε μεγάλη μας χαρά κύριε Αντιπρόεδρε. Έχετε έρθει πολλές φορές εδώ και δεν μιλάμε βέβαια για τις ακροάσεις, αλλά τα είπαμε και μετά τις ακροάσεις. Πολύ καλό αυτό. Και επίσης υπενθυμίζω ότι η Επιτροπή μας ήδη έκανε ανταλλαγή απόψεων μεσά στις 26 Ιανουαρίου του 2015 πριν εγκριθεί η στατική για την ε, ενεργειακή πολιτική. Και στην ε, Ολομέλεια του Φεβρουαρίου είχε υποβληθεί η δέσμη μέτρων για αυτή την πολιτική. Κύριε Αντιπρόεδρε, τα είπαμε ε, λίγο πριν αρχίσει η συνεδρίαση. Για μας παρουσιάσετε επομένως τα βασικά στοιχεία αυτής της ε, στρατηγικής. Όλοι γνωρίζουμε ότι η υλοποίηση είναι κάτι το πάρα πολύ βασικό, να δούμε πώς θα έχουμε καλύτερη νομοθεσία και πιο ε, αποτελεσματική. Πολύ σημαντικό σημείο αυτό για την στρατηγική. Έχουμε 15 ε, σημεία εδώ. Για να δούμε τι θα γίνει με τις σχετικές πρωτοβουλίες νομοθετικές και μη που θα αναλυθούν. Και επίσης εμείς με τη σειρά μας θα διαρθρώσουμε αντίστοιχα το έργο μας και θα δώσουμε ε, στα αντίστοιχα θέματα με εσά την προτεραιότητα. Τι σκητάρι έχετε κύριε Αντιπρόεδρε εσείς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ αγαπητέ Γέρζη. Ξιότιμοι κύριε βουλευτέ, χαίρομαι που για άλλη μια φορά ήρθα εδώ να ανταλλάξουμε απόψει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτό η Ενεργειακή Ένωση, να σα ενημερώσω για το πού βρισκόμαστε. Όπω είπε και ο Πρόεδρο, πριν από δύο μήνε συναντηθήκαμε και είπαμε στι λεπτομέρειε του τι θέλετε εσείς να περιλαμβάνει αυτή η ενεργειακή στρατηγική. Ξέρω ότι είστε ειδικοί στο θέμα, τα έχετε μελετήσει και ελπίζω ότι καλυφθήκατε. Σε ποια σημεία σας συζητήσαμε μαζί και όσα ήδη έχετε πει για την ενέργεια, για το κλίμα, ότι όλα αυτά καλύφθηκαν από την στρατηγική πλαίσιό μας. Είδατε ότι τήρησα το λόγο μου. Αυτό σημαίνει ότι άπαξ και εγκριθεί αυτή η στρατηγική πρόκειται να την παρουσιάσουμε στην Ολομέλεια. Οπότε σας ευχαριστώ για αυτή την πάρα πολύ θετική εμπειρία της συζήτησης γιατί διαπιστώσαμε το πώς οι βασικές πολιτικές ομάδες υποστηρίζουν αυτή την κοινή ευρωπαϊκή γραμμή για την ολοκληρωμένη μας πολιτική. Από τότε βέβαια δουλέψαμε πάρα πολύ ε, σκληρά με τα κράτη-μέλη, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε ότι το Συμβούλιο Ενέργειας, ε, Μεταφορών κλπ. Και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ίδιο, ότι θα υποστηρίξουν αυτή τη νέα προσέγγιση και έτσι θα ξεκινήσουμε αυτή την ε, μετάβαση στην ε, Ευρώπη ήταν πολύ σημαντική. Και την περσμένη εβδομάδα επίση οι Ευρωπαίοι ηγέτε είπαν ότι θα υποστηρίξουν πλήρω το έργο μα. Οπότε αυτό ήταν ένα μήνυμα πάρα πολύ δυνατό που είπαν ότι επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για την Ενεργειακή Ένωση επί τη βάση των προτάσεών μας και τονίστηκε το πόσο σημαντικέ είναι και οι πέντε σχετικές διαστάσεις. Οπότε είπε το Συμβούλιο πρέπει να γίνει πλήρης ε, ε, υλοποίηση και εφαρμογή αυστηρή της υπάρξης νομοθεσίας ώστε να έχουμε τα σχέδια υποδομής για να μπορεί να υπάρχει συμμόρφωση ε, για το φυσικό αέριο με όλους τους εξωτερικούς προμηθευτές. Αυτό ήταν πολύ βασικό σημείο και το είχαμε πολλές επιφυλάξεις πριν το περιλάβουμε και αυτό στην ενεργική στρατηγική. Επίσης είπαν οι ηγέτες ότι πρέπει να υπάρχουν ε, περισσότερη συνεργασία, περιφερειακή, θα πρέπει να βάθουν προσπάθειες για την αποτελεσματική της ενέργειας, για τα οικοδομήματα, επίσης για την διπλωματία σε σχέση με ε, ευρωπαϊκή διπλωματία για το κλίμα εν ώψη του COP21. Οπότε είπαμε ότι έτσι θα πρέπει να έχουμε κάποια από τα αποτελέσματα και θα έχουμε αυτούς τους βασικούς τέσσερις στόχους. Άρα πρόκειται να καταβάλουμε ε, ε, πολλή προσπάθεια ή σαν την προσπάθεια που καταβάλαμε μέχρι τώρα και όπως τα είπε ακριβώς και ο πρόεδρος Μπούζεκ. Τώρα έχουμε μια τέτοια στρατηγική και μπορέσαμε να βρούμε την κατάλληλη συνένεση. Τώρα όμως θα πρέπει αυτή η συνένεση να γίνει συγκεκριμένες ε, πράξεις, δράσεις, νομοθετικές προτάσεις, βήματα τέλος πάντων ούτω ώστε να έχουμε την σωστή συνεργασία και από δική σας πλευράς. Οπότε, αν μου επιτρέπετε, για να δούμε τώρα πώς θα ε, επισημάνουμε τους τέσσερις βασικούς στόχους. Πρώτα-πρώτα να εξασφαλίσουμε ότι για την ενεργειακή ασφάλεια η ελληνική και η εμπιστοσύνη πάβουν να είναι κενές χωρίς νόημα λέξεις. Και όλα τα ξέρουν ότι μπορούν να στηρίζονται σε κάθε περίσταση Στου γείτονέ του. Δεύτερον, θα πρέπει, όπω είπε ο πρόεδρος Γιούνκερ, να έχουμε μια πέμπτη ελευθερία. Την ελεύθερη διακίνηση της ενέργειας και να έχουμε επομένως ενεργικέ ροέ διασυνοριακά με όλους που ήρθα σε επαφή στις τελευταίες εβδομάδες από όλα τα κοινοβούλια, από όλη την Ευρώπη, με όλους τους υπεύθυνους για λήψη αφάσεων σε εθνικό επίπεδο, σε ε, τοπικό επίπεδο, με κοινωνία των πολιτών, επιχειρηματίες κλπ. Όλοι ε, μου, μου είπαν το ίδιο. Μου είπαν όλοι ότι θα πρέπει να υπάρξει μια τέτοια ελευθερία για ελεύθερη ροή της ενέργειας και έτσι να κάνει αυτό το μεγάλο προς την εμπρός η Ευρώπη προς ε, μια ολοκληρωμένη και αποκεντρωμένη ενεργειακή αγορά τρίτον. Τρίτος στόχο. θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι σκεφτόμαστε και ενεργούμε έχοντας κατά νου την αποτελεσματική χρήση της ενέργειας ακριβώς ε, όπως και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναφέρθηκε και παρέπεμψε στην αποτελεσματική χρήση της ενέργειας το οποίο άμεσα συνδέεται με το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Επομένω και σε Ευρω... επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ε, θα πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτόν τον στόχο και για όλες μας τις πολιτικές να έχουμε υπόψη το θέμα της αποτελεσματικής χρήσης της ενέργειας. Τέταρτον, να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε μια μετάβαση προς μια οικονομία με χαμηλή χρήση άνθρακα και ότι θα εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες της Ευρώπης να είμαστε ένας κόμβος για όλο τον κόσμο ούτω ώστε να έχουμε μια νέα γενιά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αυτό να γίνει με πολιτική καινοτομία και έρευνας. Έχουμε τις υποδομές που τώρα στείνονται. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε τι έγινε με το ΤΑΝΑΠ, τον αγωγό αερίου της Ανατολίας, που ξεκινά από την ε, Κασπία και ακολουθεί αυτόν τον ε, διάδρομο ε, προς τον νότο. Και έτσι θα έχουμε διαφοροποίηση όσον αφορά τις ενεργές πηγές. Επίσης έχουμε την συμφωνία Γαλλίας, Ισπανίας και Πορτογαλίας για το φυσικό αέριο και αυτό ας γίνει παράδειγμα προς μίμηση γιατί και αλλού στην Ευρώπη θα πρέπει να αναβαθμιστούν οι δυνατότητες των διασυνδέσεων. Οπότε έχουν αληθεί τώρα και δυνατικές προσπάθειες τόσο ώστε να σταθεροποιηθούν οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Την Παρασκευή προείδρευσα στις συνομιλίες Ρώσων και Ουκρανών Υπουργών Ενέργειας Συνεφώνησαν όλοι ότι θα πρέπει από τώρα να ετοιμαστούμε για την διάθεση αποθεμάτων για τον επόμενο χειμώνα του χρόνου. Επίσης, έχουν αληφθεί και ενέργειες διπλωματικές για να μπορέσουμε να έχουμε μια δεσμευτική συμφωνία και φιλόδοξη, η οποία είναι στο Παρίσι φέτος, χάρη στις προσπάθειες του Επιτρόπου Άριας Κανιέτε. Και θα είμαστε οι πρώτοι που θα αναλάβουμε αυτή τη δράση που ονομάζεται INDC, αυτή την ε, στοχευμένη και εθνικά περιχαρακωμένη συμβολή. Και έτσι θα πείσουμε και τους άλλους ε, σημαντικούς παίκτες και εμπλεκομένους, τόσο ώστε να κάνουν το ίδιο όπως και εμείς, αμελητή. Επίσης, θα πρέπει να αναλάβουμε και κάποιες νέες και πολλές πρωτοβουλίες, νομοθετικές και μη νομοθετικές. Όλος χάρη της πορείας Ένωσης για τα επόμενα πέντε χρόνια είναι αρκετά εκτεταμένος οπότε. Για να δούμε ποιες είναι πρωτοβουλίες που έχουμε τώρα εστιάσει την προσοχή μας. Έχουμε τώρα αναπτύξει το Smart Financing for Smart Buildings. Ε, ευφυής χρηματοδότηση για ευφυή ε, κτίρια. Και έτσι θα τονίσουμε το ότι όσον αφορά τα ακίνητα πρέπει κάτι να κάνουμε. Δηλαδή με κάθε τρόπο θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητές μας και σύντομα να υλοποιηθεί και να σας παρουσιάσουμε αυτή την πρωτοβουλία. Επίσης, στρατηγική για θέρμανση και ε, κλιματισμό το καλοκαίρι. Γιατί όπως είπαμε, η κρίση αφορά και την κρίση για την θέρμανση. Επίσης θα αναθεωρηθεί η οδηγία για τις ενεώσιμες πηγές ενέργειας και για την πλασματική χρήση της ενέργειας. Γιατί έχουμε τους το 2030 και φαντάζομαι θα έχουμε συγκεκριμένη πρόταση και θα σας την υποβάλουμε το 2016. Χάρη στην ε, πρόοδο που έχει στο Κοινοβούλιο η υπόθεση των αποθεματικών της ε, σταθερότητας αγοράς. Έχουμε το καινούργιο σύστημα το οποίο και αυτό έχει συμβάλει για το COP21. Ε, αυτό θα είναι μήνυμα προς την βιομηχανία να έχουμε μια ρύθμιση προβλέψιμη. Οπότε και να έχουμε ένα ETS προσαρμοσμένο αναγκές της βιομηχανίας. Επίσης να έχουμε ένα στέρεο πλαίσιο διακυβέρνησης. Ακριβώς αυτό που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τα όσα έχει δεσμευτεί να κάνει. Και να έχουμε επίση την πρωτοβουλία για την ε, πρωτοπόρα ε, ε, πολιτική της Ευρώπης όσον αφορά την καινοτομία γιατί είπαμε ότι έτσι θέλουμε να έχουμε μια ρύθμιση ε, δίκαιη και κανείς να μην είναι ουραγός γιατί χρειάζονται τώρα δεξιότητες σημαντικές για την ε, αγορά Αύριο θα έχουμε την πρώτη ε, συνεδρίαση για την στρατηγική. Και έτσι θα έχουμε τους αρμόδιους επιτρόπους για αυτές τις προτάσεις. Ελπίζουμε λοιπόν επίσης εξ αρχής ε, να μπορέσουμε να συστήσουμε μια ομάδα η οποία θα ασχοληθεί με όλα αυτά τα θέματα και θα διασφαλίσουμε να σας καταθέσουμε ποιοτικέ προτάσεις ε, για νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες τα αντικατοπτρίζουν όλα τα στοιχεία εκείνα τα οποία είναι απαραίτητα, πρέπει να ληφθούν υπόψη οποτεδήποτε προετοιμάζουμε τις νομοθετικές προτάσεις. Και γνωρίζω ότι αύριο ε, θα συζητήσετε με τον συνάδελφό μου και ξέρω ότι θα μπείτε σε περισσότερες λεπτομέρειες ως προς τις νομοθετικές προτάσεις. Θα κλείσω λοιπόν με τρία θέματα. Το πρώτο έχει σχέση με την διακυβέρνηση. Εδώ λοιπόν επιτιμούμε να προετοιμάσουμε φακέλους ε, για κάθε κράτος μέλος, ε, χαρτοφυλάκια περισσότερο, για να γνωρίζει ο καθένας ε, τι έχει να αποκομίσει, γιατί είναι σημαντική η Ενεργειακή Ένωση για τη χώρα του, γιατί πρέπει να συνεργαστεί για αυτό το project. Και αυτό το μήνυμα να το μεταφέρουμε σε πολιτικό επίπεδο, επιχειρηματικό, κοινοβουλευτικό επίπεδο, έτσι ώστε να μπορούν να ξεκινήσουν όλες αυτές οι συζητήσεις με τα κράτη-μέλη. Θα συνεργαστούμε στενά με εσά για όλες τις ε, νομοθετικές προτάσεις που αναφέρονται στον κατάλογο και επίσης ε, θα ελέγξουμε πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε τις εκθέσεις που κατατίθενται από τα κράτη-μέλη στην Κομισιόν. Θα επανέλθουμε τον Νοέμβρη και θα σας παρουσιάσουμε την πρώτη έκθεση για την ενεργειακή κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα είναι η βάση των συζητήσεών μας και θα οδηγήσει στις συζητήσεις ε, σε επίπεδο κορυφής. Γιατί πιστεύω ότι η Ενεργειακή Ένωση πρέπει να προχωρήσει σε όλα τα πολιτικά επίπεδα. Θα συνεργαστούμε στενά με την τοπική αυτοδιοίκηση. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να συνεργαστούμε σε αυτή την έννοια των ευφύων πόλεων. Ο κύριος Γιούν και ο κύριος Κατάινεν και εγώ και μια άλλη ομάδα επιτρόπων ο, Υπουργός, ο Επίτροπος Μεταφοράς και η Επίτροπος Κρέτσου όλοι αυτοί θα συνεργαστούν στενά για να παρουσιαστεί μια νέα στρατηγική για τις ευφύης πόλεις και για τις κοινότητες του μέλλοντος. Αυτά στηρίζονται όχι μόνο στην Ευρώπη όπου έχουμε πολύ καλά παραδείγματα στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη αλλά και στην Ασία και πρόσφατα και στην Αίγυπτο. Κατόπιν τούτου υπάρχει ένα σχέδιο που πρέπει να υπάρχει για Ευρώπη ευρωπαϊκές ανάγκες. Και τρίτον θα εργαστώ ακούραστα για να υπάρχει υγιής κατάσταση ενέργειας... στην κεντρική και τη νότια Ευρώπη. Είναι το πρόγραμμα ΚΕΣΕΚ, αφορά την σύνδεση αυτού του τμήματος της Ευρώπης με το υπόλοιπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οφείλουμε να διασφαλίσουμε κάθε μία από αυτές τις χώρες να έχουν τη δυνατότητα σε παροχή αερίου τουλάχιστον από τρεις διαφορετικές πηγές. Πρέπει να βοηθήσουμε αυτή την περιοχή να ενταχθεί καλύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό μπορούμε να το κάνουμε σε στενή συνεργασία ε, ε, με ε, χώρες που συμμετέχουν <coughs> ήδη ε, στη διαδικασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταλλαγή απόψεων που αφορούν στην Ενεργειακή Ένωση. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συνεισφορά σας, για τη βελτίωση της στρατηγικής και προσβλέπω στην περαιτέρω συνεργασία, γιατί θεωρώ ότι κάτι τέτοιο θα είναι απολύτως απαραίτητο. Και εμείς ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε και ξεκινάνε οι συζητήσεις. Πρώτος γύρος ερωτήσεων, οι συντονιστές. Παρακαλώ, όχι περισσότερο από τρία λεπτά ο καθένας. Το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, σας ε, χαιρετίζω κύριε Αντιπρόεδρε και θέλω να σας πω και συγχαρητήρια διότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου πράγματι είναι ε, ουσιαστικά και από ό,τι φαίνεται υπάρχει και στήριξη των κρατών μελών για τη σύσταση της Ενεργειακής Ένωσης. Ε, δεν ξέρω αν το έχετε μπροστά σας, αλλά θέλω να σας επισημάνω το ΔΕΛΤΑ, το D των συμπερασμάτων, όπου το Συμβούλιο αναφέρει ότι θέλουν να διασφαλίσουν την πλήρη συμβατότητα με το κοινοτικό δίκαιο, αυτό ε, για τις νομοθετικές ρυθμίσεις ε, και όχι μόνο για να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και συμβατότητα με τις ε, κοινοτικέ διατάξεις. Και αυτό αφορά την παροχή αερίου. Εκεί είναι σημαντική και η εχεμήθεια. Ξέρω ότι αυτό το δούλεψε πολύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την τελευταία θητεία για να υπάρχει πιο ενεργός ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, σε διαπραγματεύσεις για κλείσιμο συμβολών με τρίτες χώρες. Τώρα το Συμβούλιο μοιάζει να μετακινείται περισσότερο στη θέση της Επιτροπής. Και θέλω να ρωτήσω, κατά τη δική σας άποψη, ε, πόσο θα προχωρήσει το Συμβούλιο. Γιατί είναι κάτι τελείως διαφορετικό να λέει θέλουμε μεγαλύτερη διαφάνεια, αλλά είναι και κάτι τελείως διαφορετικό να ε, υπάρχουν κοινά στοιχεία σε όλες τις διαπραγματεύσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας επ' αυτού. Ο κύριος ε, Ντανίκα από τους ε, Σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα μιλήσω ε, ρουμάνικα επειδή έχω την ευκαιρία να μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα. Και θα ήθελα ε, κύριε Αντιπρόεδρε να σας ε, συγχαρώ για αυτά που μας είπατε. Μας παρουσιάσατε επικαιροποιημένη την κατάσταση και επίσης είπατε ότι οι συζητήσεις για την Ενεργειακή Ένωση στην Ευρώπη είναι σημαντικές και ότι τώρα υπάρχει και ένα σαφές χρονοδιάγραμμα. Οι τιμές για τους καταναλωτές και για τους χρήστες είναι πολύ σημαντικές και εξαρτώνται και από εύρυθμα λειτουργούσες αγορές. Πώς θα πείσετε τις επιχειρήσεις για τη χρησιμότητα της Ενεργειακής Ένωσης. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια κοινή αγορά. Αυτό θα είναι πιο αποτελεσματικό και θα μειωθούν οι τιμές. Όσον αφορά τις ενεργειακές υποδομές, η, ε, τα σημεία σύνδεσης θα πρέπει να χρηματοδοτούν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και χαίρομαι για αυτά που είπατε για τον Νότιο Διάδρομο και για την Κασπία γιατί κατά το παρελθόν δεν ήταν σαφές πώς μπορούμε να επιτύχουμε την αποτελεσματικότητα. Το θέμα είναι ότι είμαστε αναγκασμένοι να εισάγουμε ε, αέριο από τη Ρωσία και τώρα αυτές οι, ε, θα κατασκευαστούν αυτές οι γραμμές διασύνδεσης, τα interconnectors. Αν λοιπόν έχουμε τέτοιες γραμμές διασύνδεσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας που είναι το 10%. Παραδείγματο χάρη την προηγούμενη εβδομάδα έγινε λόγος για τα solar clips και βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια ε, ευαίσθητα τμήματα, κάποια θέματα που δεν έχουν ολοκληρωθεί. Ε, γιατί σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε ότι χάθηκαν πολλά μεγαβάτ, υπήρξαν διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος και ήταν θαύματο ότι αποφύγαμε blackout στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να γίνουν ε, σε αυτό το επίπεδο. Βεβαίως Αύριο ε, μπορούμε να μιλήσουμε και για ένα πολύ σημαντικό θέμα, αλλά όσον αφορά τις ε, γραμμές διασύνδεσης, ε, θα το μοιραστείτε το θέμα με τον κύριο Καγέτη ή πώς θα το μοιράσετε. Και όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, πώς θα μοιράσετε τις αρμοδιότητες ανάμεσά σας γιατί δεν είμαστε σίγουροι ε, με ποιον θα πρέπει να έρθουμε σε επαφή αν υπάρξουν προβλήματα. Μήπως μπορείτε να μας ενημερώσετε. Σας ευχαριστούμε για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζετε την νέα αγορά στην Ευρώπη. Επόμενος. Σας ευχαριστούμε και τώρα ε, ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη κύριε Επίτροπε. Είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργεία θα πρέπει να έχει ως σκοπό τη μεγαλύτερη ασφάλεια, την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ο σκοπό έχει να αυξήσει και την ασφάλεια αλλά και την εμπιστοσύνη στο σύστημα. Θα ήθελα να μας εξηγήσετε κύριε Επιτροπέ τι ακριβώς εννοείται με τον όρο αυτό. Μιλάμε για την εμπιστοσύνη που έχουμε ένα τον άλλον, αλλά σε ό,τι αφορά την Ενεργειακή Ένωση. Έχουμε και το θέμα της ε, χρήσης και της έκκλησης λιγότερου άνθρακα. Τι γίνεται λοιπόν με τον άνθρακα ως ενεργειακό πόρο. Αν θέλουμε πιο ασφαλή, πιο υγιεινά και περιβαλλοντικά λιγότερο επιβαρυντικά συστήματα για την παραγωγή ενέργειας, τι γίνεται με τον άνθρακα. Αυτό δεν αφορά μόνο τα στρατηγικά συμφέροντα της χώρας μας, της Πολωνίας, αλλά και την άμεση απειλή της βάρος της ενεργειακής ασφάλειας, γιατί αν ε, είναι να είμαστε όλο και πιο εξαρτημένοι από παρόχους ενέργειας, δεν είμαι βέβαιος ότι αυτό κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Έχετε, λοιπόν, κύριε Επίτροπε, τον αντίκτυπο στην Πολωνία αλλά και σε άλλες χώρες όπου η κατάσταση είναι παρόμοια και κοιτώντας ε, πως έχει η κατάσταση σε ό,τι αφορά την ε, ενέργεια και την παροχή ενέργειας, βλέπουμε ότι δεν εφαρμόζεται η αρχή ε, της μη διακριτικής μεταχείρισης ύστερα σε ό,τι αφορά το αέριο, τι γίνεται. Τρίτο ζήτημα σε ό,τι αφορά ένα μηχανισμό κρίσης, ε, σε ό,τι αφορά τους μηχανισμούς και τους χώρους αποθήκευσης. Στη συνέχεια, σε ό,τι αφορά το οικονομικό και νομικό πλαίσιο, σε ό,τι αφορά τις μη συμβατικές ε, πηγές ενέργειας, όπως μέσω της συντροδογμάτωσης τι γίνεται, κατά πέμπτον. Προτείνεται μια ριζοσπαστική πραγματικά διαφοροποίηση των προμηθευτών μια τέτοια ενεργειακή ένωση δεν παρέχει όμως δυνατότητες πραγματικής γρήγορης ανάπτυξης για χώρες όπως η Πολωνία. Και μακροπρόθεσμα θα είμαστε όλο και πιο εξαρτημένοι από τις εισαγωγές ανέργειας. Τι γίνεται λοιπόν κύριε Επίτροπε σε ό,τι αφορά την αρχή της εμπιστοσύνης και της αλληλεγγύης όπου ακούμε πολλές και διαφορετικές απόψεις. Για να συνοψίσω, Αυτά που προβλέπει το Συμβούλιο για τους διάφορους ενεργειακούς φορείς και για την χρήση λιγότερου άνθρακα στην ε, ενέργεια σε συνδυασμό και με την ατζέντα για το κλίμα. Ίσως θα έπρεπε να αλλάξουμε το όνομα και τον τίτλο της, του εγγράφου και να μην είναι η Ενεργειακή Ένωση μόνο το θέμα, αλλά και η κλιματική πολιτική, γιατί ουσιαστικά μια πολιτική για το κλίμα ασκούμε και χώρες όπως ε, και η Γερμανία. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα από την άλλη έχουμε τον ε, επόμενο μελητή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τον Αντιπρόεδρο Σεύκοβιτς ε, για τη σκληρή δουλειά που έκανε και που μας δίνει την ευκαιρία να συζητήσουμε και πάλι μαζί εδώ στην Επιτροπή μας. Αυτό καταδεικνύει πόσο μεγάλη είναι πραγματικά η δέσμευσή του για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Θα ήθελα να θίξω δύο βασικά ζητήματα για την ομάδα της ΑΛΔΕ. Το θέμα της διακυβέρνησης και το θέμα της χρηματοδότησης. Ακούω τα σχόλιά σας και τις σκέψεις σας για εκθέσεις ανά χώρα. Η, ιδέα να υπάρχει μια αιτήσια κατάσταση και απολογισμός, αν θέλετε, της Ενεργειακής Ένωσης, μου φαίνεται ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα για να συζητιόνται τα βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε. Όλοι ξέρουμε ότι το ενεργειακό μείγμα αποτελεί, σύμφωνα με τις εθνικές, εθνική αρμοδιότητα και εκ παραλλήλου προφανώς χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη ενεργειακή αγορά που θα επιτρέπει μεγαλύτερη διασύνδεση για να υπάρχει μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια και για να υπάρχουν και πιο πολλέ ανανεώσιμες στο ενεργειακό δίκτυο. Και παρά την αντίφαση αυτή βλέπουμε ότι υπάρχει πρόοδος στη διασύνδεση, στο επίπεδο διασύνδεσης και χαίρομαι που υπάρχει μια σωστή εξέλιξη από πλευρά των συμπερασμάτων του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά το 10% σε επίπεδο στόχο κτλ. Θα ήθελα να ακούσω όμως ποιες είναι οι δικές σας σκέψεις κύριε Αντιπρόεδρε για το βασικό αυτό το δίλημα και τις συζητήσεις που γίνονται μέσα στο Συμβούλιο σε σχέση με το τι αποτελεί η εθνική κυριαρχία και το πώς μπορούμε από κοινού να ενισχύσουμε την Ενεργειακή Ένωση. Και επίσης, για να αναπτύξτε μας λίγο αυτά που αναφέρω από το... στα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την πλήρη εφαρμογή το... της ήδη φυστάμενης ενεργειακής νομοθεσίας. Τέλος παράθεση. Τι σημαίνει αυτό. Έχει να κάνει με τις εκθέσεις αναχώρα. Σας παρακαλώ, για πείτε μας λίγο παραπάνω. Και τέλος μία ερώτηση για τη χρηματοδότηση. Το έχω θέσει και στο παρελθόν το ερώτημα αυτό. Σε ό,τι αφορά έργα κοινή ωφέλεια, κοινού συμφέροντο, πόσα τέτοια έργα είναι σε φάση που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι σχεδόν βιώσιμα για χρηματοδότηση, πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα σημαντικά έργα θα πάρουν την χρηματοδότηση που χρειάζονται και μπορούν να προχωρήσουν. Και τέλος, πώς θα συμπεριλάβουμε έργα για την ενεργειακή αποδοτικότητα στο πλαίσιο αυτό. Θα ήθελα πραγματικά να ακούσω το σχόλιο που έχετε να κάνετε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος ε, συνάδελφος Τούρμες, από τους Πράσινους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ και εσάς, Αντιπρόεδρε Σεφκοβίτς, εσείς και η ομάδα σας ε, στην Επιτροπή Κάνετε πραγματικά πολύ καλή δουλειά. Δεν μας ικανοποιούν όλα, αλλά υπάρχουν καλά σημεία για την πλήρη εφαρμογή του 2020 για να, για διασφαλίσουμε ότι η αποδοτικότητα με τη νέα νομοθεσία θα είναι στο επίκεντρο. Επίσης, το ότι καταλαβαίνουμε επιτέλους ότι η κρίση με τη Ρωσία είναι θέμα θέρμανσης και ότι λαμβάνουμε πρωτοβουλίες και επίσης πρώτη φορά δίνεται ένας ρόλος στους, στις ευρωπαϊκές πόλεις. Κρίσιμο ζήτημα αυτό. Χρειάζεται τέτοιου είδους πρόοδος και επίση. για τις περιφέρειες τι ε, αγορές τις μικροπεριφερειακές που είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, ένα ζήτημα το οποίο είναι αντιφατικό ασφαλώς. Έχω τρεις, ε, τρία, τρία σημεία. Καταρχάς, καλή κίνηση προς την διαφάνεια για το φυσικό αέριο στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Αλλά για μένα ανακύπτει το ερώτημα τι θα κάνουμε με μια χώρα όπως η Ουγγαρία. Μια χώρα που για διάφορους λόγους κινείται εντελώς αντίθετα προς την αλληλεγγύη των άλλων. Με ό,τι διαφάνεια και να έχουμε, σε τελική ανάλυση θα πρέπει να δράσουμε αν κάποιος είναι αντίθετος με τα συμφέροντα της Ευνεργειακής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, ελεύθερη ροή και παροχή ηλεκτρισμού. Πολύ ωραία ιδέα. Αλλά αν είναι σε μια τελείως στρεβλωμένη αγορά αυτή η ελεύθερη παροχή ηλεκτρισμού, όπου δεν υπάρχει σωστή τιμολόγηση, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πολύ περίεργες αποφάσεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διεξάγει μία μελέτη για τις κρατικές επιδοτήσεις. Τα αρκετά καύσιμα είναι πρώτα, δεύτερον τα πληνικά και τρίτον οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Χθες το απόγευμα, μάλλον Παρασκευή, Σάββατο, η γερμανική κυβέρνηση σε επίσημη μελέτη του Υπουργείου ε, ομολόγησε ότι η Γερμανία δεν έχει αρκετά χρήματα για να αποχαρακτηρίσει τους πυρηνικούς αντιδραστήρες. Τι κάνουμε λοιπόν, αποδεχόμαστε ότι οι φορολογούμενοι τελικά θα πληρώσουν εκατοντάδες, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ίσως και όχι οι διαχειριστές των αντιδραστήρων αυτών. Αυτό αποτελεί μία από τις πιο τεράστιες στρεβλώσεις. Το 2003 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε υποσχεθεί να προτείνει ένα ταμείο για τον σωστό καταμερισμό των έξοδων από χαρακτηρισμό. Τι κάνατε λοιπόν, τέλος, στο θέμα τη σωστή και έξυπνη χρηματοδότηση για έξυπνα κτίρια. Smart financing for smart buildings. Μάλιστα. Αλλά όταν αποφασιστεί το OFC δεν θα έχουμε άλλα χρήματα. Δεν θα έχουμε άλλα κονδύλια. Ελπίζω λοιπόν από το σύστημα το Smart Financing for Smart Buildings να υποστηρίξει την ενεργειακή αποφαντικότητα που θα προκαλέσει περίπου 50 δισεκατομμύρια και βάλε επενδύσεις, γνωρίζοντας ότι έχουμε τέτοιο τεράστιο κενό στην χρηματοδότηση της ε, ανανέωσης και της, ε, των κτηρίων. Σε ό,τι αφορά την έκλειψη τώρα, την ηλιακή έκπληξη, ήμουν στο Βερολίνο την ε, Παρασκευή Εκατοντάδε χιλιάδε άνθρωποι είχαν ξεχυθεί στου δρόμου. Και φυσικά ο γερμανικό τύπο, γιατί είχε γίνει φυσικά μεγάλη... Είχαν γίνει πολλές εικασίες και υποθέσεις για blackout κτλ. Στον 2 λοιπόν το απόγευμα μίλησα με πρόσωπο της γερμανικής κυβέρνησης και μου είπε ότι για δεύτερη φορά στη ζωή μου έφτασα στο αμήν. Γιατί το δεκαετία του 80 ε, είχε χρειαστεί να τεθεί ένα θέμα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των πυρηνικών αντιδραστηρίων στη Γερμανία. Τότε δεν είχε συμβεί τίποτα. Όλες αυτές τις ιστορίες λοιπόν μου είπε για το σύστημα ηλεκτροδότησης το οποίο δεν θα ανταπεξέλθει υποτίθεται στις ε, συνθήκε, Κατά τη γνώμη του εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία. Αυτό λοιπόν που έγινε την τελευταία Παρασκευή την προηγούμενη Παρασκευή καταδεικνύει ότι είναι μια χαρά τα συστήματά μα, Έτοιμα να αντιμετωπίσουν τέτοιε προκλήσεις. Ο κ. Ελικιώτη τώρα από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, και εγώ θέλω να, να συγχαρώ τον Αντιπρόεδρο ε, και για τη δουλειά που γίνεται η ομάδα του παρόλο που ε, έχουμε και εμεί σημαντικέ ε, διαφωνίες και διαφορετικέ απόψει. Βεβαίω, βέβαια να συγχαρώ γιατί ε, με τη συχνή του παρουσία εδώ στην Επιτροπή Φαίνεται να αντιλαμβάνετε τη σχέση που πρέπει να υπάρχει μεταξύ του ε, Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Ε, δεν θα αναφερθώ σε θέματα που τα είπαμε και άλλες φορές ε, και κυρίως τη διαφωνία μας για την ενισχυμένη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε διακρατικές, σε διακρατικές συμφωνίες και στις διαπραγματεύσεις ενώ όσο υπάρχει ακόμα και δεν βλέπουμε να υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα για την άρση της απομόνωσης κρατών και περιοχών. Ούτε είμαστε ικανοποιημένοι με τις προτάσεις που έχει να κάνει με την ενεργειακή φτώχεια. Και εγώ θα ξεκινήσω με δύο ζητήματα που α, α, τίθενται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το πρώτο είναι να αφορά για την ανάγκη διασφάλισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών κατά την εξερεύνηση και ανάπτυξη των φυσικών του σπόρων. Και εδώ ε, έχουμε ένα κράτος μέλος όπως είναι η Κυπριακή Δημοκρατία που προχωρά σε αυτές τις ενέργειες και όμως βλέπουμε ε, να υπάρχουν παράνομες ε, ενέργειες από πλευρά της Τουρκίας, μια υποψήφια προσένταξη χρόνα, να παρενοχλεί το κράτος με πλοία και παρόλα αυτά στην ανακοίνωση περιλαμβάνεται μια πολύ θετική αναφορά στην Τουρκία και στο ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η την ενεργειακή ασφάλεια παραβλέποντα αυτόν το γεγονό τη παραμπόδοση κρατών μελών από το να ασκήσουν τα κυριαρχικά του δικαιώματα όπω εκφράζονται και στα συμπεράσματα. Το δεύτερο είναι ακόμα μια αναφορά που υπάρχει στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι το ζήτημα της αξιοποίησης των εγχώριων πηγών. Και όμως κύριε Αντιπρόεδρε, ε, το ξαναείπα σε τέτοιες εδώ και κατά την ακρόαση σα και με άλλες ευκαιρίες, θεωρώ ότι ε, και μέσα από αυτήν την ανακοίνωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση παραβλέπονται πρώτα-πρώτα ε, ε, ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει και η Κύπρος αλλά και ευρύτερα τα κοιτάσματα στην Ανατολική Μεσόγειο για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ένωσης. Και μάλιστα σε μια στιγμή που ήδη υπάρχει παραγωγή φυσικού αερίου ε, ε, από κοιτάσματα στην περιοχή και αναφέρομαι στα κοιτάσματα του Ισραήλ. Ήδη πριν από λίγες μέρες η Αμερικανική εταιρεία Ενόπολ που ε, έχει τα δικαιώματα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου προχωρά σε λίγες εβδομάδες να κηρύξει εμπορεύσιμο το κοίτασμα και γίνεται ένα πρόγραμμα ανάπτυξης. Άρα περνούμε πλέον από το στάδιο της έρευνας στο στάδιο της ανάπτυξης. Ε, και στην Κύπρο όπως βεβαίως και στην ευρύτερη περιοχή. Ε, και ε, εδώ ακριβώς είναι το ερώτημα μα ποιες είναι οι σκέψεις της Επιτροπής μέσα στα πλαίσια της στήριξης της ενεργειακής ασφάλειας αυτά τα σημαντικά κοιτάσματα που βρίσκονται και σε έναν κράτο αλλά και σε μια περιοχή που συνορεύει με την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως είναι η Ανατολική Μεσόγειο. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ντάριο Ταμπουράνο από το EFTD, παρακαλώ, έχει το λόγο. Αυτά που είπατε ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα και πράγματι είναι σημαντικό να υπάρχει μεγαλύτερη διασύνδεση ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Εμείς θεωρούμε ε, ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι επιτέλους ε, κατέστη σαφές ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διασύνδεση ανάμεσα στα ηλεκτρικά δίκτυα. Ε, ήδη αυτό τη δεκαετία του 80 ελέγχθη από τον κύριο Φούλουρ. Ε, πέρασαν 30 χρόνια, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Βεβαίως ε, θέλω να πω ότι αυτή η Ενεργειακή Ένωση θα βασίζεται στα εθνικά μονοπόλια και θα είναι το πλεονέκτημα των μεγάλων γραμμών διασύνδεσης ενώ μέχρι τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν μικρά κράτη και μικρά χωριά ακόμα και μικρές περιφέρειες που δεν μπορούν ε, καν να ανταλλάξουν μεταξύ τους ηλεκτρικό ρεύμα, ηλεκτρική ενέργεια. Άρα δηλαδή στην Ιταλία τουλάχιστον ε, σημαίνει αυτό. Ε, πρέπει να σκεπτούμε και μακρο ενεργειακά αλλά και μικροενεργειακά που αφορά τα χωριά, την τοπική αυτοδιοίκηση. Όχι να δώσουμε πλεονέκτημα μόνο στις πόλεις και να έχουμε μόνο κατά νου τις ευφύης πόλεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και κύριε Αντιπρόεδρε για όλα αυτά που μας είπατε σήμερα. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω για τις ε, προσπάθειες που καταβάλατε τις τελευταίες εβδομάδες για να παρουσιάσετε θέματα ενεργειακής ένωσης. Θα ήθελα να εξετάσω ένα συγκεκριμένο θέμα, το οποίο δείξατε κι εσείς στον τομέα της Ενεργειακής Ένωσης θα ήθελα να ασχοληθούμε με τα πυρηνικά, όχι τόσο με την έρευνα και την ανταγωνιστικότητα. Εσείς ο ίδιος είπατε ότι κυρίως όσον αφορά τη μετάβαση ε, σε μια Ενεργειακή Ένωση χαμηλής ε, κατανάλωσης άνθρακα είναι σημαντικό για να γίνει αυτό να είναι πιο ανταγωνιστική η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και σε επίπεδο επιχειρήσεων και σε επίπεδο ανανόσιμων πηγών ενέργειας. Να υπάρχουν δηλαδή επενδύσεις με σημαντική υπεραξία και αυτό που ενδιαφέρει είναι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να επικρατήσουν σε διεθνές επίπεδο να υπάρχουν συγκεκριμένες αλυσίδες παροχής ενέργειας. Επίσης, στήξατε και το θέμα των κρατικών προμηθειών ε, και εκεί πρέπει να ληφθεί υπόψη η πράσινη ανάπτυξη. Νομίζω ότι έτσι μπορούν να προκύψουν ε, τεχνολογίες κλειδί. Είπατε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να έχει μια πολυτομεακή προσέγγιση. Και ρωτώ, υπάρχει χρονικό πλαίσιο για αυτή την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα στοιχεία που να μπορείτε να μας καταθέσετε ήδη σήμερα. Και δεύτερον, όσον αφορά τη χρηματοδότηση αυτής της ε, πρωτοβουλίας, ε, Ίσως μπορείτε να μας ενημερώσετε λιγάκι για το πώς ε, τελικά θα χρηματοδοτηθεί αυτή η πρωτοβουλία. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Αντιπρόεδρο για να απαντήσει. Στο πρώτο γύρο των ερωτήσεων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Για τόσα είπατε και για τόσα ρωτήσατε. Και τον κύριο Κάρινς. Είναι πολύ θετικό το ότι και εσείς ε, έτσι βλέπετε όπως και εγώ, τις αποφάσεις του Συμβουλίου σαν μια πολύ σημαντική πολιτική κίνηση. Πριν από λίγα χρόνια είχαμε ομόφωνη υποστήριξη για να έχουμε περισσότερη διαφάνεια για τα IGA και επίσης για τη συμβάση του ιδιωτικού τομέα. Κάτι το οποίο ήταν δύσκολο κανείς το παρελθόν να το σεβαστεί, να το φανταστεί. Οπότε Είπαμε ότι και με τη συζήτηση στο Κοινοβούλιο τονίστηκε το πόσο σημαντική υπόθεση είναι η διαφάνεια και επίσης το πόσο σημαντικό πολιτικό εργαλείο είναι αυτό που έχουμε στα χέρια μας. Και αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να έχουμε δίκαιες συνθήκες στην ευρωπαϊκή αγορά. ποιότητα, πληροφορίες, ακριβώς όπως και στην άλλη πλευρά του τραπεζιού με αυτούς με τους οποίους διαπραγματευόμαστε. Γιατί πολλές φορές υπήρχαν πληροφορίες αλλά δεν μας τις έλεγαν. Ή τις διαφορές τις τιμολογιακές τι πληρώνει κάθε χώρα το φυσικό αέριο. Αυτές όλες οι συνθήκες που ήταν τόσο δύσκολο να ξεπεραστούν. Γι' αυτό και λέω ότι η διαφάνεια είναι κάτι το πολύ καλό. Είναι η ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτήν τόσο άνηση κατάσταση. Αυτό θέλω να δούμε το πώς θα υλοποιηθεί. Ακριβώς όπως έλεγε ο κύριος Κάρινς και ρώτησε σχετικά τώρα δούμε θα γίνουμε αυτές τις δύο προτάσεις. Πρώτα-πρώτα η απόφαση για τις ε, διακυβερνητικές συμφωνίες. Να υπάρχει εκ των προτέρων έλεγχος και όχι εκ των υστέρων ο έλεγχος για αυτές τις συμφωνίες. Και πίστηκαν τελικά οι αρχικοί κρατών και κυβερνήσεων και οι αρμόδιοι υπουργοί. Ας πούμε για το South Stream. Διαπραγματεύσεις, κύρος των συνθήκων, αλλά είδαν ότι δεν συνάδουν προς το κοινοτικό δίκαιο. Οπότε είχαμε ένα σωρό προβλήματα. Άρα είπαμε να μην ξεχνάμε τα ίδια λάθη όπως το παρελθόν. Οπότε είπαμε στην διαπραγματευτική ομάδα να έχουμε τους ε, νομικούς μας, να υπάρχει επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να έχουμε κάποιες κοινέ ρήτρε και να εξασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε τέτοιου συμφωνία θα αφιγραμμίζεται με την κοινοτική νομοθεσία. Και αυτό θα είναι καλό για τα κράτη-μέλη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για όλους τους οικονομικούς παράγοντες που θέλουν να μπορούν να βασιστούν σε αυτές τις ε, συμφωνίες ε, να έχουν κάποια σταθερότητα να βασιστούν. Τώρα, για τη συμβάση του τομέα και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να δούμε πώς θα αναθεωρήσουμε την οδηγία για το φυσικό αέριο. Να δούμε τι έγινε πέρσι, ε, να δούμε πώς θα γίνει πιο ανθεκτικό το σύστημα. Οπότε και οι εταιρείε μας και τα κράτη-μέλη να μπορούν να έχουν ένα περιβάλλον αξιόπιστο στο οποίο να κινηθούν. Ξέρουμε τι θα πει εμπιστευτικές πληροφορίες. Αλλά οι πληροφορίες αυτές για, το, για τα benchmark και όλες αυτές οι πληροφορίες οι εμπιστευτικές είναι πολύ χρήσιμες στις εταιρείε. Και επίσης η Ευρώπη μπορεί πια να είναι πιο ισχυρό διαπραγματευτής όταν υπάρχει αυτή η πληροφόρηση για όλους κατόπιν δεν υπήρχε μέχρι σήμερα. Και έτσι, με την νομοθεσία που θα θεσπίσουμε, θα μπορούσαμε να πείσουμε τους υπουργούς, τα κρατημέλη, τις ε, εταιρείε για την κατεύθυνση που θέλουμε να πάρουμε. Ένας άλλος ε, κύριος ε, ρώτησε κάτι σχετικά με τις τιμές και θεώρησα ότι αυτό είναι πάρα πολύ βασική ένδειξη για το αν πάμε καλά για την Ενεργειακή Ένωση. Να υπάρχει νεωνιστικό περιβάλλον, και έτσι να υπάρχει συμπίεση των τιμών προς τα κάτω. Αυτό είναι και θέμα υποδομών. Θα πρέπει να καλύψουμε το έλλειμμα που έχουμε και επίσης θεωρήσα πολύ θετικό το ότι υπάρχει ε, θετική απόκριση από την ε, Νότια Ευρώπη. Δεν θα πρέπει να κολλάμε στα πολύ μεγάλα προγράμματα και έργα. Μην θεωρούμε ότι αυτά θα λύσουν όλα μας τα προβλήματα. Να δούμε τι γίνεται με τις διασυνδέσεις, με τα ε, μικρότερα προγράμματα και έργα. Αυτά θα μας δώσουν ολοκλήρωση, θα μας δώσουν διασυνδεσιμότητα. <coughs> και έτσι θα εξασφαλίσουμε τον έχουν αυτές οι χώρες επιλογές και πρόσβαση στην ενέργεια. Και όταν είπαμε κυρία Πέτκοβα την Υπουργό Ενέργεια τη Βουλγαρία και μου εξήγησε το ότι η Βουλγαρία σημαίνει πρόοδο σε όλα τα μέτωπα για τι διασυνδέσει, όπω χρειάζεται η χώρα. Τελευταίου μήνε τα πράγματα κάπω έχουν κολλήσει, αλλά και τώρα βλέπουμε να υπάρχει κινητικότητα. Γι' αυτό το 10% και για το αν θα μπορούσαμε να το υλοποιήσουμε, είπαμε ότι 12 κρατημέλη είναι κάτω από αυτό το όριο αυτό το στόχο του 10% αλλά μέχρι το 2020 όλα τα μέλη εκτός από την Κύπρο θα έχουν πετύχει το στόχο αυτό. Υπάρχει όμως ο ευρωασιατικός διασυνδετικός, ε, διασυνδετικός για την ε, Κύπρο. Οπότε θα έχει 100% διασυνδεσιμότητα η Κύπρος. Ελπίζουμε ότι αυτό το έργο θα βρει την αναγκαία υποστήριξη. Και εάν μπορέσουμε να υλοποιήσουμε όλα τα PCI, αυτά τα οποία προτείνουμε εμείς, ελπίζουμε να έχουμε πετύχει όλοι το 10% και οπότε πια ο πύχης να ανέβει για το 2030. Τώρα για να δούμε δύο διαπραγματεύσει. Ο επικεφαλής των προτεύσεων για την Επιτροπή είναι ο Άρια Κανιέτε. Συνεργαζόμαστε πολύ στενά. Δουλεύουμε ομαδικά και επίσης θα συνεργαστούμε με τον Κανιέτη και την Φεντερίνη Μογκερίνη, τον Επιτροποχάν και έτσι οι διπλωματικές αυτές προσπάθειες ελπίζουμε να πείσουν τις χώρες που πρέπει ούτως ώστε και αυτές να συμμετάσχουν στις έννοιες που απαιτείται στις διαμονητεύσεις του COP21. Και έτσι πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε κάποια συμφωνία που θα δεσμεύει όπως θέλουμε. Ο κ. Γιάνκεβης τώρα είπε τι θα γίνει με την ενεργειακή ασφάλεια για τις αγορές φυσικού αερίου και άνθρακα. Θα συζητήσετε εδώ Επιτροπή σας τι γίνεται με την ε, αγορά, που θεωρείτε ότι λειτουργεί εύρυθμα και ότι δεν χρειάζεται περαιτέρω βελτιώσεις. Όμως αυτά είναι στη Δυτική Ευρώπη, στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Οπότε χρειάζεται μια προσέγγιση αυτή που προτείνουμε να μελετήσει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα πράγματα και σύντομα θα φανεί πώς έχουν τα πράγματα και πώς μπορούμε να έχουμε και εκεί κάποια κατάλληλα μέσα πολιτικής που να συνάδουν προς τις δεσμεύσεις μας των ΠΟΕ. Και οπότε μέσα στη συγκυρία της κρίσης να μπορέσει να διπλωματευτεί όπως χρειάζεται η Ευρώπη και έτσι να αντιμετωπίσει την κρίση. Επίσης, διάφοροι βουλευτές ε, είχαν κάποια θέματα εθνικής κυριαρχίας σε σχέση με τις ε, ε, εθνικές αρμοδιότητες και τους στόχους τους ενεργειακούς. Έχουμε τις κυρίαρχες αποφάσεις για την ενέργεια, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να σεβαστούμε το πλαίσιο το οποίο μαζί το αποφασίσαμε. Και με τα άλλα μείγματα πολιτικής θα πρέπει να φτάσουμε και να πετύχουμε τον στόχο μας για το κλίμα. Νομίζω ότι έχουμε καλύψει την αφετηρία μας ε, και γι' αυτό και ήταν ομόφωνη η απόφαση του Οκτωβρίου. Ε, και τελικά προσχώρησε σε αυτήν και η Πολωνία. Πιο γρήγορα θέλετε να τα πω κύριε Πρόεδρε. Ε, very telegraphic. I will be very, very telegraphic. Uh, Mr. Peterson was asking about... κύριος Πέτερσεν για τα PCI και την βελτιωμένη διακυβέρνηση. Οπότε τώρα θα πρέπει να δούμε πώς θα χρηματοδοτήσουμε αυτά τα PCI. Έχουμε ε, το Green Euro έχουμε τα διευθυντικά ταμεία, σύντομα θα έχουμε το στρατηγικό πλάνο Juncker, οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η διακυβέρνηση, οπότε και αυτή η τρεις αγωγοί του προγράμματος θα κατατείνουν σε έναν στόχο. Και όσον αφορά τις υποδομές και έτσι θα καλύψουμε την, ε, τις προτεραιότητές μας. Ακριβώς όπως έχουμε πει. Για το EFCI. Βελτιωμένη διακυβέρνηση. Και έτσι θα εξασφαλίσουμε το ότι θα κάνουμε τα κατάλληλα διαβήματα. Κύριε Τούρμες, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και τις προτάσεις για το μέλλον. Αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό για αυτά τα οποία συστήσατε είναι το να δούμε πώς θα μπορούμε να έχουμε μια καινούργια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Άρα χρειάζονται κάποιες προτάσεις για το μέλλον. Αν λοιπόν σχεδιάζουμε σωστά την αγορά, όλα αυτά δεν τα σχετικά με τις επιδοτήσεις όσον αφορά την εμπλοκή στα σύνορα, ε, όλα αυτά που θα λυθούν με αυτή την προσέγγιση. Ο κύριος Σιλικιώτης και ο κύριος Ταμπουράνο αναφερθήκατε στην ε, ενεργειακή φτώχεια και τα σχετικά ζητήματα. Ε, συνεργάζομαι με την κυρία Τάισεν και με τα κρατημέρια για να πώ θα μπορούσαμε να έχουμε τα κατάλληλα μέσα πολιτική, κοινωνική πολιτική, για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτού που δεν μπορούν να πληρώσουν την ακριβή ενέργεια. Και για τον κύριο Σιλικιώτη επίση, ε, να τον ενημερώσω ότι για την θέματα της εθνικής κυριαρχίας και τα δικαιώματα εκμετάλλευσης από τα κράτη-μέλη είναι κατηγορηματικό το Συμβούλιο στα συμπεράσματά του. Όπως είπατε και κάποια άλλη βουλευτή που είπε για ε, καινοτομία, έρευνα, χρηματοδότηση πολιτικών και γι' αυτό είπαμε ότι οι πράσινες πολιτικές θα περάσουν σε όλο τον ε, προϋπολογισμό. και επομένως να διοπτρίζεται αυτή μας η γραμμή σε όλα τα προγράμματα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θα προτείνω, θα προτείνω να κλείσουμε τον κατάλογο των ομιλητών. Δεν βλέπω να ζητάει κανείς άλλο το λόγο. Να κλείσουμε τον κατάλογο των ομιλητών, αλλά 1,5 λεπτό αναμιλητή. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Η κυρία Φαμπρέντ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως ξέρετε κύριε Αντιπρόεδρε, και εμείς ως ομάδα στο Κοινοβούλιο καλωσορίζουμε ιδιαίτερα στην Ενεργειακή Ένωση. Δεν είναι σημαντικό ασφαλώς κάθε μέτρο ξεχωριστά όσο το σύνολο, το άθροισμα των μέτρων. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να πω ότι είμαι μάλλον ευχαριστημένη με τη συμφωνία του Συμβουλίου παρά το γεγονός ότι όλοι γνωρίζουμε ότι χρειάστηκαν διπλωματική λιγμή ε, για να τα αποτύχουμε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, καλό όμω είναι και ήδη καταδεικνύει μια αλλαγή νοοτροπία και το γεγονό ότι υπάρχει Ενεργειακή Ένωση, το γεγονό ότι υπάρχει ολιστική προσέγγιση σε ό,τι αφορά την ενέργεια και το κλίμα, αυτό είναι καθοριστικό. Μπορούμε να κάνουμε μια εξελιτική συζήτηση για την ενεργειακό μείγμα, αν και νομίζω ότι είναι σημαντικό το θέμα αυτό, ας επικεντρωθούμε σε αυτά που συμφωνούμε, σε αυτά που μας βρίσκουν σύμφωνος. Ενεργειακή αποδοτικότητα πρώτη και καλύτερη, το είπατε και εσείς. Και είπατε και κάτι πολύ σημαντικό στο πλαίσιο αυτό, το θέμα των εφιών πόλεων. Τα μικρά έργα που έχουν να κάνουν και με την ενέργεια αλλά και με τη διασύνδεση του ψηφιακού κόσμου. Να ενώσουμε τα θέματα της Ενεργειακής Ένωσης και της ε, ψηφιακής διασύνδεσης. Το θέμα του ΕΦΣΙ, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και συζητιέται ιδιαίτερα στο Κοινοβούλιο, πρέπει να δείξουμε ανοιχτό χαρακτήρα. Όταν μιλάμε για επενδύσεις σκεφτόμαστε αεροδρόμια, δρόμους, αυτοκινητόδρομους και εκεί χρειάζεται μια διαφορετική νοοτροπία και εδώ μπορούμε να διασυνδέσουμε την Ενεργειακή Ένωση. Και φυσικά και χρειάζονται τα μεγάλα έργα, αλλά η Ενεργειακή Ένωση έχει να κάνει και με τα μικρά project και με τις ευθύνες πόλεις. Ξέρετε ότι θα ήθελα να τα... Ήθελα να ρωτήσω, ο Πρόεδρος παραμένει, Πώ θα θέλετε να το πετύχετε αυτό. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Επόμενος ομιλητή, η κυρία Βέρνερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, να σα συγχαρώ κι εγώ για την στρατηγική πλαίσιο και κυρίω για την ταχύτητα που προχωράτε και ελπίζω να συνεχίσετε να προχωράτε με τόσο γρήγορους ρυθμούς, να έχουμε γρήγορα προτάσεις από την Ενεργική Ένωση. Δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις, γιατί δεν έχω και χρόνο. Μου προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι στον οδικό χάρτη για την ε, Ενεργειακή Ένωση, στο 3α, αναφέρεται ότι η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που πρόκειται να δημοσιεύσει για την ε, πυρηνική ενέργεια, η Euratom, η συνθήκη, υποχρεώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημοσιεύει στοιχεία τακτικά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι μάλλον ατυχές, θεωρώ, και σε ό,τι αφορά την χρονική συγκυρία και σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες να μπαίνει αυτό ως τμήμα της Ενεργειακής Ένωσης, ένα τμήμα δηλαδή για την πυρηνική πολιτική, γιατί με την Ενεργειακή Ένωση αυτό που θέλουμε να πετύχουμε, έτσι καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον, είναι μια ενεργειακή παραγωγή και ένα γεγικό μοντέλο φιλικό προς το περιβάλλον. Θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε ποια είναι η τοποθέτησή σας για την προτεραιότητα αυτή. Και δεύτερη ερώτηση σε ό,τι αφορά αυτό που είπε ο Κλοντ Τούρμες, αυτή η μελλοντική αγορά ηλεκτρισμού στην Ευρώπη. Θα δημοσιεύσει σχετικό πρόγραμμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέτο και του χρόνου νομοθετική πρόταση. Θα μπορούσατε να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω γιατί μιλάμε και για την ενίσχυση της ενία Ευρωπαϊκή αγοράς άλλωστε. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα ο κύριος Γκέρικα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ενεργειακή αποδοτικότητα Αποτερεί το σκληρό πυρήνα της Ενεργειακής Ένωσης. Τώρα έχουμε πραγματικά εργαλεία και για τον κλάδο αλλά και για τα μεμονωμένα κρατημέλη γιατί ο τρέχον στόχος του 40% είναι πολιτικής φύσεως και έχει να κάνει με περιορισμούς ως επιτοπλίστων. Η τρέχουσα οδηγία, και εδώ είμαι αντίθετος με την κύριο δεν έχει αποδείξει ότι είναι χειρότερη. Το μοναδικό εργαλείο για την αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να είναι η τελική αποδοτικότητά της. Και η κατάσταση διαφέρει σε πολλά γιατί σε θέματα παραγωγής και κατανάλωσης. Αλλά οι προτάσεις αυτές δεν προωθούν την καινοτομία σε ό,τι αφορά θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας, ούτε τις ανανεώσιμες. Πώς θα λάβετε λοιπόν υπόψη το κενό αυτό την έλλειψη αυτού του εργαλείου στο ETS. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Ζωρίνιο είναι επόμενος ευχαριστώ, Κύριε Αντιπρόεδρο, να σας συγχαρώ που κάνετε αυτή τη συζήτηση για την Ενεργειακή Ένωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό καταδεικνύει τον ενθουσιασμό και την ε, ορμή που υπάρχει. Είναι σημαντικό λοιπόν να τα αξιοποιήσουμε αυτά και να προωθηθούν οι καθαρέ πηγέ ενέργεια και η καταπολέμηση τη ενεργειακής ένδυας. Εκ παραλλήλου θα πρέπει να μειώσουμε τα απορρίμματά, μα τα και την άσκοπη σπατάλη ενέργεια. Δύο ερωτήσεις έχω να σα κάνω. Καταρχά την προτεραιότητα που δίνεται στις ανανεώσιμες. Σωστή και δίκαιη. Παρ' όλα αυτά, μπαίνει στο πλαίσιο της ε, προοπτικής της αγοράς. Οι ανανεώσιμες θα πρέπει να είναι ανταγωνιστικές στην αγορά, θα πρέπει να έχουν ανταγωνιστικές τιμές. Πολύ σημαντικό αυτό. Σε ό,τι αφορά την Ενεργειακή Ένωση, θα πρέπει καταρχάς να προβλεφθεί ένα εργαλείο το οποίο θα ενισχύσει την έρευνα και την ανάπτυξη. Για τους λόγους αυτούς ακριβώς. Αν θέλουμε να παράγουμε ανανεώσιμη ενέργεια από ανανεώσιμε πηγέ θα πρέπει να υπάρχει ανταγωνιστική τιμή στην αγορά. Δεν έχει νόημα να πωλείται η ενέργεια αυτή στην αγορά με μη ανταγωνιστικέ τιμέ όπω γίνεται στη χώρα μου και σημαντικό επίση είναι να μην στραβλώνει τον ανταγωνισμό ο οποίο υφίσταται στην αγορά, κοιτώντα για παράδειγμα το συστολεκτικό αέριο στη ΣΥΠΑ και σε άλλα μέρη του κόσμου. Βλέπουμε ότι γίνεται παραγωγή σχιστολιθικού αερίου και εγώ ο ίδιος τήρτησα μία έκθεση για το συστηλικωτικό αέριο συζητήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο Παναμά. Και φαίνεται ότι γίνονται πολλές αναφορές στο συστολιτικό αέριο στις διάφορες συμφωνίες, παρά το γεγονός ότι δεν αποτελεί ακόμα προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση η στρατηγική αυτή για το συστολιτικό αέριο, σίγουρα θα αποτελέσει σημαντική μορφή ενέργειας και θα πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική λοιπόν από πλευρά μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριο Πίπερ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Αντιπρόεδρο καταρχήν για την ενεργειακή επάρκεια. Είπατε ότι πολλά πρέπει να εκτιμιστούν από μόνο του στην αγορά. Η τελευταία όμω ενεργειακή οδηγία διευκολύνει την κατάσταση και λέει δεν θα ασχοληθούμε με την αποτελεσματικότητα αλλά με την εξοικονόμηση. Κάθε χρόνο, κάθε κράτο μέλο ε, πρέπει να εξοικονομήσει 1%. Και το ερώτημά μου είναι, εσείς ε, πώς θα προχωρήσετε σε αυτήν την ενεργειακή επάρκεια. Δηλαδή θα πείτε κι εσείς ότι θα επιβάλλουμε εξοικονόμηση ή μήπως αυτή τη φορά θα υπάρχει κάποια μεγαλύτερη ευελιξία. Το δεύτερο ερώτημα που θέλω να σας κάνω αφορά ε, τις ε, αγορές δυναμικού. Δηλαδή κάθε χώρα εξετάζει αυτό το θέμα του δυναμικού. Εσείς ε, πώς προτίθεστε αυτές τις ε, διαφορετικές ε, εξελίξεις που υπάρχουν στη Γαλλία, στη Γερμανία να τις εντάξετε σε ένα και μόνο ολοκληρωμένο πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σεφκοβίτς για το γεγονός ότι έρχεται τόσο συχνά στην Επιτροπή μας και επιδεικνύει τέτοια επιμέλεια ε, και συνέπεια ε, στην παρουσία του στη συναντήση μας. Αυτό αποδεικνύει από μόνο του το πόση σημασία αποδίδουμε στην ενέργεια. Ε, είμαι ευγνώμων για την παρουσία του και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική. Επίσης συμφωνώ με την προσπάθεια που καταβάλλεται να συσταθεί κοινή αγορά. Ε, θα έπρεπε να συσταθεί και δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Ένα από τα βασικά θέματα είναι η υποστήριξη της, ε, των δυνατοτήτων διασύνδεσης. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Υπάρχει όμως κάτι το οποίο αντιβαίνει ε, αυτήν την προσπάθεια, δηλαδή το πώς ακριβώς προσεγγίζουμε το θέμα των ε, επιδοτήσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που πολλές φορές ε, είναι μακροπρόθεσμες και μακροχρόνιες. Πώς θα το αντιμετωπίσει το θέμα, γιατί τελικά υπάρχει κίνδυνος να αλλάξουν τα συμβόλαια αναδρομικά που μπορεί να σημαίνει διαιτησία, ε, μπορεί να σημαίνει ε, μακροχρόνιες διενέξεις. Θέλετε λιγάκι να μας ενημερώσετε πάνω σε αυτό. Παρακαλώ, ο κύριος Αντιπρόεδρος έχει το λόγο. Α, ο κύριος Μπιτικόφερ. Ε, κύριε Αντιπρόεδρε, δεν θέλω τώρα να σας επιδεψιλεύσω φιλοφρονήσεις. Υπάρχει χρόνος για αργότερα για κάτι τέτοιο. Έχω κάποιες ε, άλλες πιο κρίσιμες παρατηρήσεις. Δηλαδή στο θέμα της ενεργικής ανεξάρτησης θα πρέπει να υπογραμμίσουμε περισσότερο ότι η αποτελεσματικότητα, η ενεργειακή και ενώσιμες πηγές ενέργειας είναι ο πυρήνας της στρατηγική μας. Και δεύτερον αυτό που θέλω να επικρίνω είναι ότι στα συμπεράσματα του Συμβουλίου ε, έχει καθοριστεί και προβλεφθεί η αρχή της ομοφωνίας όπου αναφέρεται ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, θα συνεχίσει να δίνει Δηλαδή αν επιθυμούμε ενεργειακή ένωση δεν μπορούμε να επιλέξουμε μια στρατηγική που θα λέω ότι ο αργότερος θα καθορίζει το ρυθμό. Όσον αφορά τώρα τη διαφάνεια για τα συμβόλαια αερίου. Ε, το συζητήξατε προηγουμένως και θα ήθελα να διευκρινίσετε κάτι τι ακριβώς, ποια, ποια, ποιο είδου συμβόλαια θα συνάπτονται. Θα είναι ανάμεσα σε κράτη, ανάμεσα σε κράτη και ιδιώτες ή αναφέρεστε σε κάθε είδου συμβόλαιο. Η κυρία Κομπολανάσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλοί μίλησαν για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και είδα λιγάκι και τα στοιχεία της Κομισιόν για τις ανανεώσιμες πηγές και η Εστονία, Βουλγαρία και η Σουηδία έχουν ήδη εκπληρώσει τους στόχους τους. Εγώ προέρχομαι από τη Φινλανδία αυτή τη στιγμή από το 38% εμείς επιτυγχάνουμε το 34,5%. Η Σουηδία και η Λετωνία είναι μπροστά. Όλοι οι άλλοι υπολείπονται ε, και πολλές από τις χώρες ασχολούνται και με τη βιοενέργεια. Θα ήθελα λοιπόν κύριε Σεύκοβιτς ή δυνατόν να μας ενημερώσετε λιγάκι για μια συνεπή πολιτική. Έχουμε πολλούς στόχους. Ε, κατά την άποψή σας ε, ποια είναι η καλύτερη χρήση της ε, βιομάζας στον, σε, για θέματα ενέργειας. Παρακαλώ κύριε Αντιπρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω ό,τι μπορώ για να είμαι σύντομος. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω την κυρία Φανμπραντ για την υποστήριξή της και επίσης ε, και αυτό που είπε θα το υιοθετήσω και εγώ ε, γιατί παρουσιάζει μια πολύ ωραία εικόνα ε, να <laughs> έχουμε δηλαδή μια κοινότητα του ήλιου και του αέρα και νομίζω ότι έτσι μπορούμε να εξηγήσουμε τις θεμελιώδεις αλλαγές που μπορούμε να επιτύχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλες αυτές οι θετικές εξελίξεις θα την χάνουν πλήρους χρήσης. Η ενεργειακή επάρκεια, η ευφυείς πόλεις, αυτά πρέπει να είναι απόσπαστα συστατικά μελλοντικών προτάσεών μας. Και συμφωνώ πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να φτάσουμε στις, ε, στους μικρούς δήμους και μικρές κοινότητες να κάνουμε περισσότερα για την ενεργειακή επάρκεια. Αυτό που μας φοβίζουν είναι οι οικονομικές πιέσεις. Ίσως να μην έχουμε ε, την διοικητική στήριξη για τέτοιου είδους προγράμματα. Αυτό λοιπόν που θέλουμε να κάνουμε είναι να μιλήσουμε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Επενδύσεων για το πώς μπορεί κανείς να ε, ολοκληρώσει αυτά τα μικρά προγράμματα και να προσφέρει απλά εργαλεία. Γιατί όταν μιλάμε με θεσμικούς επενδυτές, κυρίως με τα συνταξιωτικά ταμεία, όλοι αυτοί θέλουν να επενδύσουν, αλλά βεβαίως θα ήθελα να δουν πώς ακριβώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο το οποίο ε, δεν θα έχει να κάνει με εκατοντάδες επίδοξους επενδυτές, αλλά να μπορούν οι μικρές πόλεις να εντάσσονται σε αυτό το δίκτυο. Και αυτό είναι ένα σημαντικό καθήκον και το καλό είναι ότι έχουμε ήδη ξεκινήσει τις εσωτερικές μας συζητήσεις με τον τραπεζικό τομέα. Όσον αφορά τώρα ε, σε αυτό που ερώτησε η κυρία Βέρνερ, κοιτάξτε όταν πρόκειται για την πυρηνική ενέργεια το θέμα είναι ότι τώρα έχουμε 16 ε, κράτη-μέλη τα οποία παράγουν ενέργεια ε, πυρηνική και κάποια εξ αυτών αποφάσισαν ότι θέλουν να συνεχίσουν. Γνωρίζω ότι εδώ έχουμε ένα πολύ σημαντικό καθήκον να διασφαλίσουμε ότι αυτό πρέπει να γίνεται με απόλυτη ασφάλεια και επίσης και ε, τηρώντας ε, τα περιβαλλοντικά πρότυπα. Άρα δηλαδή πρέπει να εξτάσουμε όλα αυτά κατά από το πρίσμα ε, των περιβαλλοντικών προτύπων. Νομίζω ότι αυτό είναι μεγάλη ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτό είναι ένα πρωταρχικό καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα, η ερώτηση του κυρίου Γκίρεκ. νομίζω αν μιλήσει κανείς με επιχειρήσεις ε, θα κατανοήσει ότι επικρατεί η άποψη αυτό που επιθυμούμε είναι η ρυθμιστική σταθερότητα. Θέλουμε να ξέρουμε ε, ποιες είναι οι αρχές της αγοράς. Οι μηχανισμοί εκείνοι που ε, θα επιτρέψουν να καθορίζουμε μια καλή τιμή άνθρακα. Άρα δηλαδή πρέπει όλα αυτά να τα διορθώσουμε, να λειτουργούν και πάλι και αυτό ακριβώς θα προτείνουμε όταν θα καταθέσουμε τη μεταρρύθμιση του ε, Ευρωπαϊκού ε, Συστήματος Ανταλλαγών. Ε, θεωρώ ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε πολλές καινοτόμες απόψεις και αυτή θα είναι και η μεταρρύθμιση που θα επιβάλλουμε. Ε, υπογραμμίστηκε η σημασία της έρευνας και της καινοτομίας. Συμφωνώ μαζί του. Ένας από τους τομείς όπου μπορούμε να επενδύσουμε περισσότερο στην έρευνα και την καινοτομία είναι πώς μπορούμε ε, να προωθήσουμε αυτά που είμαστε ήδη ισχυροί, όπως τα ευφυή e e δείγματα και ευφυή e πλαίσια. Ε, μπορούμε να πείσουμε τους ε, καταναλωτές ότι αυτοί θα αποφασίζουν για τα ενεργειακά πλέγματα ε, και να είμαστε σίγουροι ότι η ενέργεια θα χρησιμοποιείται με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από ό,τι σήμερα ίσως να μην υπάρξει μια επανάσταση με το σχιστόλιθο όπως στις Ηνωμένε Πολιτείε. Μπορούμε όμως να έχουμε μια επανάσταση σχετικά με τα ενεργειακά πλέγματα. Αυτό ε, αρέσει πολύ στους νέους που χρησιμοποιούν όλα αυτά τα FEE κινητά, τα smartphones. Ε, μπορούμε να διεκδικήσουμε παρεμφερή αποτελέσματα και θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε σε αυτό και την υποστήριξή σας. Ο κύριος Πάιπερ ρώτησε ε, τι θα κάνουμε με την ενεργειακή επάρκεια. Νομίζω είναι απόλυτα σαφές ότι ε, θα πρέπει να ανανεώσουμε την οδηγία για την ενεργειακή επάρκεια, επίσης την οδηγία για τα κτίρια ε, και όλα αυτά είναι πολύ συγκεκριμένες προτάσεις τις οποίες πολύ σύντομα θα συζητήσουμε ε, βεβαίως ε, προηγουμένως ε, θα έχουμε διαβουλέψεις, γιατί αυτή τη φορά θέλουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, πιο στοχευμένοι και με τον τρόπο αυτό πιστεύουμε ότι θα παρουσιάσουμε καλύτερα αποτελέσματα. Όσον αφορά τώρα το δυναμικό των αγορών Νομίζω ότι αυτό ε, σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας νέος σχεδιασμός. Συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να επιτύχουμε καλύτερα οικονομίες κλίμακος και σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο. Έχουμε το φόρουμ των ε, χωρών της Βαλτικής με τις ε, σκανδιναβικές χώρες και αυτοί μας δείχνουν πόσο αποτελεσματικός μπορεί να είναι κανείς αν συνεργάζεται σε ε, περιφερειακό επίπεδο. Επίσης ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο που κάνατε ότι έρχομαι εδώ συχνά και με επιμέλεια προσπαθώ να μη μακρηγορώ, να είμαι λακωνικός αλλά συμφωνώ μαζί σας ότι για να υπάρχει κοινή αγορά είναι καθοριστική σημασία η διασύνδεση όπως και η άρση εμποδίων που ε, μας, ε, δεν μας βοηθούν στο να επιτύχουμε καλές ενεργειακές τιμές. Για την αναδρομικότητα ε, και τις διάφορες αριθμίες που έχουμε στις ενεργειακές αγορές. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εφαρμόσουμε οδηγίες για τις κρατικές ενισχύσεις, τις παρουσιάσαμε πέρυσι, για τις ε, ανώσιμες πηγές ενέργειας, για το περιβάλλον και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλα αυτά θα λειτουργούν στο ίδιο επίπεδο ανταγωνιστικότητας και επίσης θεωρώ ότι έτσι ε, θα έχουμε και πολύ καλύτερες αναλύσεις. Ας δούμε λιγάκι ποιες είναι οι ενεργειακές δομές στην Ευρώπη. Γιατί υπάρχουν αυτές οι τιμές ε, της ε, χονδρικής ε, που μοιάζει με αυτές που υπάρχουν στις ΗΠΑ αλλά είναι τελείως εδώ διαφορετική η τελική τιμή διότι περιλαμβάνουμε ε, διαφορετικά φορολογικά συστήματα, πολλά τέλη και εισφορές άρα δηλαδή πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τον τελικό καθορισμό των ενεργειακών τιμών στην Ευρώπη. Ο κύριος Πίτικοφερ επισήμανε το θέμα της ενεργειακής επάρκειας και το ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε με κάποια ανωνυμία. Αυτό ε, είναι πολύ σημαντικό, έτσι ίσχυε πάντα. Βεβαίως όσον αφορά τις ε, νομοθετικές προτάσεις υπάρχουν οι κλασικές ε, προτάσεις όπου συμπεριλαμβάνονται οι κανονικές και εκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρώ ότι μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ετέθηκε ένα ερώτημα σχετικά με τα συμβόλαια. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει όλες οι διατάξεις να είναι συμβατές με τις διατάξεις μας, δηλαδή διαφάνεια για όλα τα συμβόλαια και όπως σας είπα προηγουμένως δουλεύουμε πάνω σε αυτό επεξεργαζόμαστε νομοθετικές ε, προτάσεις ε, που έχουν και σχέση προφανώς με την προμήθεια φυσικού αερίου. Η τελευταία ερώτηση είναι από την κυρία Κούπλα Νούτρη για τη βιομάζα. Νομίζω η βιομάζα είναι πολύ σημαντική πηγή ενέργειας. Σουηδία, Φιλανδία και χώρες της Βαλτικής ε, μπορούν να αλλάξουν το ενεργειακό τους σκηνικό ε, και να ανεξαρτητοποιηθούν ε, χρησιμοποιώντας τους πόρους με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η ενεργειακή στρατηγική, λέει ο Πρόεδρος, είναι ένα από τα βασικότερα θέματα της δικής μας της Επιτροπής και θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας αύριο το απόγευμα στις 3 η ώρα με τον κύριο Κανιέτε που θα είναι κοντά μας και επίσης ε, θα προετοιμάσουμε και τη δική μας έκθεση για τη Στρατηγική Ένωση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Colleagues, ladies and gentlemen, let us go forward. Ε, συνάδελφοι, ας συνεχίσουμε. Ναι. Δεν έχουμε λεπτό να χάσουμε. Too spoiled. Uh, point number five in our agenda. Στο 5 της ημερήσιας διάταξης έχουμε τη διάδοση γεωσκοπικών δορυφορικών δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς. Συνάδελφοι, λέω, καθίστε. Wouldn't like to be together with us, so sorry to move Όσοι δεν να μείνουν για τη συζήτηση, να βγουν γρήγορα και ήσυχα. Thank you to all of you uh, Συνάδελφοι, διάδοση γεωσκοπικών δορυφορικών δεδομένων για εμπορικού σκοπούς. Όπως ξέρετε, σκοπός της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να δημιουργήσει μία εσωτερική αγορά για δορυφορικά δεδομένα. Η Επιτροπή ΙΜΚΟ διασυνδεδεμένη βάση του κανόνα 54 μαζί με τη δική μας Επιτροπή. Και έγινε και πρόταση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πολύ σημαντικό αυτό για μα, να αποσυρθεί η πρόταση αυτή, αν δεν μπορούσε να βρεθεί συμφωνία εντό έξι μηνών μεταξύ της πρόταση, ε, μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Αλλά ο πρώτος αντιπρόεδρος κ. Τίμερμαντς ανακοίνωσε στις 10 Μαρτίου στην ε, διάσκεψη των επικεφαλής ε, των Επιτροπών α, ότι η Επιτροπή δεν πρόκειται να αποσύρει την πρόταση εφόσον ε, συνέχισαν να δουλεύουν επ' αυτής και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Η κυρία Κρέλ είναι η συγγήτριά μας. Σας παρακαλώ. Πάρτε το λόγο και παρουσιάστε μας την έκθεση αυτή. Πέντε λεπτά, όχι παραπάνω σας παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόκειται δεν πρόκειται για την έκθεση ακόμα, πρόκειται για ναι, έγγραφο εργασία. Φαντάζομαι ότι πολλοί συνάδελφοι κρίνουν ότι είναι πιο σημαντική η Ενεργειακή Ένωση από τα δορυφορικά δεδομένα. Αλλά σε κάποια χρόνια θα είναι διαφορετικά τα πράγματα, ναι. γιατί είμαι απόλυτα πεπισμένη ότι ο διαστημικός τομέας αποτελεί ένα κατεξοχή τομέα για την έρευνα και την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την στρατηγική για το 2020 έχει μεγάλο ρόλο για την βιώσιμη οικονομία. Τα δορυφαρικά προϊόντα και οι υπηρεσίες που κατίστανται είναι όλο και πιο σημαντικά για τους πολίτες και, τις Ευρωπα... και την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να το αντιλαμβάνονται απόρριτα για παράλληλα επικοινωνίες. Πρόγνωση καιρού Αυτά είναι γνωστά σε πολλούς, αλλά άλλοι τομείς ε, που επηρεάζονται πολεοδομία, γεωργία, τηλεπικοινωνίες, ε, παρακολούθηση, γεωπαρακολούθηση. Όλα αυτά αποτελούν βασικούς πυλώνες ε, της διαστημικής πολιτικής. Άρα για την οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι καθοριστικό να υπάρχει το σωστό κανονιστικό πλαίσιο για να υπάρχει και η σωστή εξέλιξη και πρόεδρος. Για να προλυάνει λοιπόν το έδαφος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη το 2013 είχε αποφασίσει να προτείνει και να δημιουργήσει ένα συνεκτικό πλαίσιο και μία, ένας έλεγχος από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχε ως αποτέλεσμα ότι ιδιαίτερα σε θέματα γεωπαρακολούθησης και για τη διάδοση και παραγωγή δεδομένων των ε, διαστημικών σταθμών ε, υπήρχε ανάγκη για μεγαλύτερο συντονισμό γιατί δεν μπορούσε να υπάρξει επαρκή συντονισμό μόνο με τι εθνικέ νομοθεσίε. Τον Ιούνιο του 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι λοιπόν κατέθεσε πρόταση οδηγία στην οποία και σκοπεύουμε να τροποποιήσουμε με την έκθεσή μας η Επιτροπή ΙΜΚΟ, η Επιτροπή ΙΤΡΕ, οι οποίες όπως είπατε κύριε Πρόεδρε σύμφωνα με το άρθρο 54 είναι διασυνδεδεμένες, ήταν στενή συνεργασία από την αρχή, προκειμένου να είναι επικοδομητική και κοινή τελικά η έκθεση. Το έγγραφο εργασίας το οποίο έχετε στη διάθεσή σας ε, το κατήρτισα με τη βοήθεια του συναδέλφου Νίλσεν για το σχέδιο οδηγίας. Σκοπός της οδηγίας είναι να δημιουργήσει μια νέα αγορά για τα δεδομένα αυτά για την πρόσβαση στην αγορά, στη διάθεση στην αγορά ε, δορυφορικών στοιχείων. Θα πρέπει να υπάρχουν κοινά πρότυπα για τη διαφάνεια, την ίση αντιμετώπιση για τα δεδομένα που προκύπτουν από τα, τα γεωσκοπικά αυτά δεδομένα για να διασφαλιστεί ότι οι εμπορικοί πάροχοι στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να διαδίδουν τα δεδομένα αυτά χωρίς ε, εμπόδια σε ό,τι αφορά τα δεδομένα τα οποία είναι σχετικά μέχρι 2,5 μέτρα για να διασφαλίσουμε και την πλευρά της ασφάλειας. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει αυτή η δυνατότητα για την ελεύθερη αγορά και πρόσβαση στην αγορά, να υπάρχει ισότητα πρόσβασης για όλους. Επιπλέον θα πρέπει η οικονομική ανάπτυξη των επιχειρήσεων να προωθείται και ενδεχόμενη διάδοση σε άλλους τομείς και να παρακολουθείτε. Πιστεύω λοιπόν ότι η προτινόμενη οδηγία έχει το δυναμικό να πετύχει τους στόχους αυτούς και ότι η οδηγία μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική επιτύχη ε, και να απευθυνθεί σε κάποια σημαντικά θέματα του διαστημικού αυτού τομέα. Κάναμε διάφορες διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς και κατά την ανάλυση της τρέχουσας πρότασης Πρέπει να πούμε ωστόσο ότι πιστεύουμε ότι υπάρχουν και κάποια προβλήματα σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τη μελέτη αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, ε, όπου ήταν πολύ λίγοι αυτοί οι φορείς και ποιοτική ανάλυση της οδηγίας ή ανεπαρκής ε, ε, ανάλυση κόστους ωφέλους. Ένα σημαντικό άλλο θέμα είναι ποια προβλήματα θα μπορούσαν να επιληθούν με την οδηγία αυτή και δεν μας ικανοποιεί ε, παρκώς η μελετή αντικτύπου που περιλαμβάνεται στην οδηγία, ούτε μας ικανοποιούν ακριβώς ε, οι αναλύσεις των προβλημάτων και το πώς μπορούν να επιληθούν αυτά τα προβλήματα. Εδώ θέλουμε λοιπόν να γίνει μια συζήτηση επί της αρχής. Αναγκαστικά θα γίνει αυτό. Παρ' όλα αυτά θα θέλαμε με τον κανονισμό αυτό, με τη ρύθμιση του κλάδου αυτού, να υπάρχει θετικό αντίκτυπο και για άλλου τομεί, όπω η γεωργία, η ναυτιπλοεία, η παραγωγή καυσίμων. Όλοι αυτοί οι κλάδοι να μπορέσουν να επωφεληθούν από μια τέτοια κοινή οδηγία. Ωστόσο, να προσέξουμε, γιατί το γραφειοκρατικό κόστος θα πρέπει να περιοριστεί για τις επιχειρήσεις. Και φυσικά θα πρέπει να λεφθεί υπόψη και η εθνική ασφάλεια η εκάστοτε. Γι' αυτό λοιπόν θα θέλαμε στην έκθεση αυτή να αναφερθούν κάποιες σκέψεις για το πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Θεωρούμε ότι σε κάποια σημεία θα πρέπει να υπάρχει πιο σαφής ορισμός για να μην είναι διαφορετικές ερμηνείες της οδηγίας, να υπάρχουν σαφείς κανόνες για όλους και σκεφτόμαστε να μπει και μια ειδική ρήτρα αναθεώρησης, γιατί ασφαλώς πρόκειται και μια, για μια ταχύτητα αναπτυσσόμενη αγορά, ένα ταχύτητα αναπτυσσόμενο κλάδο και θα πρέπει να μπορούμε να προσαρμοζόμαστε. Αυτά με μια υπέρβαση του χρόνου ομιλίας για αυτό το θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον συναρπαστικό, αλλά νομίζω ότι έχουμε και χρόνο να το συζητήσουμε με τους συναδέλφους. Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ε, έχετε δίκιο, είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψη για το θέμα αυτό. Και έχουμε όλη τη διαδικασία που τώρα ξεκινάει και θα συζητήσουμε και και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει τώρα είναι η σειρά των ε, σκιωδών εισηγητών. Ο κ. και είναι ο πρώτος αγωρητής. Πρόεδρε, ευχαριστώ και συμφωνώ με τον εισηγητή μας την συγγήτριά μας, συγγνώμη, και να την ευχαριστήσω γιατί πάρα πολύ ε, εύστοχα τα είπε και πάρα πολύ λογικά. Θα πρέπει να μην ξεχνούμε το πόσο σημαντικά είναι τα συστήματα τα οποία έχει η Ευρώπη. Επίσης, θα πρέπει να μην ξεχνούμε ότι η Ευρώπη δεν είναι η μόνη κοινότητα κρατών που έχει πρόσβαση σε τέτοια υψηλή τεχνολογία. Επομένως, θα πρέπει να υπάρξει ένα νομοθετικό, κανονιστικό πλαίσιο, αν μη τι άλλο για λόγους ασφάλειας. Και αν είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, βέβαια να μην στρεβλώσουμε την αγορά, διότι αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να συμβεί. οι φωτογραφίες αλλά γενικότερα και τα δεδομένα που προέρχονται από τους δορυφόρους θα μπορούσαν να λάβουν άλλες κατευθύνσεις. Θα μπορούσαν να είναι επίσης φραγμός στην ε, βιομηχανία και στις επιχειρήσεις. Να κάτσουμε και να ε, ζυγίσουμε επομένω τις επιπτώσεις. Να δούμε ακριβώς τι πάμε να κάνουμε με αυτή τη ρύθμιση. η ασφάλεια είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι το βασικό επιχείρημα που αφορά αυτή τη συζήτηση για τους κανονισμούς που θέλουμε να θεσπίσουμε. Εν πάση περιπτώσει προσβλέπουμε στην ε, συνεργασία με τη συγκήτρια και θεωρούμε ότι πρόκειται για πολύ σημαντική έκθεση και θα αποτελέσει προηγούμενο για το πώς θα ρυθμίσουμε όλες τις τεχνολογίες που έχουν επιπτώσεις στην ενεργειακή ένωση. Άρα μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δώσουμε στο θέμα. Ο επόμενος. Ε, κυρία Κόρμαν Νιόεν Χιούτον, συγγνώμη αν δεν μου πρόφερα καλά το όνομά σας. Σας γνωρίζω, εν πάση περιπτώσει ξέρω ότι περί ημών πρόκειται. Όχι, όχι, το είπατε σχεδόν ε, τέλεια, λέει η κυρία Νιούν Χάουζεν Βίμπεγκα. Μέχρι τώρα τα πήγα πάρα πολύ καλά με την εισηγήτρια της. Τα συζητήσαμε και την ευχαριστούμε για την πρωτοβουλία της. Πάντως, όπως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει πρώτα-πρώτα να, αναρωτηθούμε τι πρόβλημα πάμε να επιλύσουμε. Χρειαζόμαστε αυτό το νομοθέτημα. Πολλά ερωτήματα ανέκυψαν. όπως ξέρετε και εσείς όταν κάνει συναντήσει τους εμπλεκομένους ε, μετά τη συζήτηση έχει πιο πολλά ερωτήματα στο μυαλό του από όσα είχε πριν. Οπότε θα πρέπει να τα δούμε τα πράγματα στις λεπτομεριές τους. Εντελεχέστερα. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε μήπως στρεβλώσουμε την αγορά όπως είχα και ο προλαλής σας. Τι γίνεται με τους δορυφόρους, ε, τους κινέζικους και τους αμερικανικούς. Τι έτσι συνέβη με αυτούς. Τι έγινε επίσης και με το διοικητικό αυτός. Θεωρήθηκε ότι θα, πρόκειται για έναν, ε, θα, για έναν φραγμό γιατί θα δημιουργήσει πολύ γραφειοκρατία, πολύ διοικητικό αυτός. Άρα, να ξαναδούμε το θέμα. Χρειάζεται να θεσπίσουμε αυτό το νομοθέτημα. Όπως έχει σήμερα η πρόταση τα κράτη-μέλη πρέπει να ορίσουν μια αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση, για τον έλεγχο όλων των εικόνων των δορυφορικών και έχουν ένα σωρό, υποχρέωση, υποχρεώσεις ε, αναφοράς και κοινοποίησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό να δούμε χρειάζεται ή ου. Πάντως ήταν πολύ σωστό ότι ξεκινήσαμε με την συνάντηση των ε, εμπλεκομένων. Οι επαφές μας ήταν πάρα πολύ επικοδομητικές, οπότε και προσβλέπουμε στην περαιτέρω συνεργασία και εμείς. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Λέω Πρόεδρος. Και τώρα. Ο κύριος Γκονσάλες έχει το λόγο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν έχουμε πολλά να πούμε σε αυτή τη φάση. Και διαπιστώσαμε ότι υπάρχει πρόθεση συνεργασίας και δεν είναι δική μου δουλειά να σας πω κατά πόσον όλα μέχρι τώρα γίνουν τέλεια. Πάντως, για να πάει καλά αυτή η πρόταση, εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και θα συνεργαστούμε όσο μπορούμε καλύτερα με το Κοινοβούλιο για να ξεκαθαριστούν κάποια πράγματα. Αυτά που πρέπει να διευκρινιστούν και όπου χρειάζεται να δουλέψουμε για να κάνουμε τις τυχόν συμπληρώσεις που χρειάζεται. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις παρατηρήσεις. Τώρα, η συγγετρία, κυρία Κρέλ. Θέλει να δευτερολογήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το είπατε και εσείς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκέφτηκε να αποσύρει την πρόταση για την οδηγία, αποφάσισε διαφορετικά, το ζήτησε άλλωστε και το Κοινοβούλιο και όντως στις 25, 25 Μαρτίου θα συνεδριάσουν τα κράτη-μέλη. Έχουν διαφορετικές απόψεις ενδεχομένως, αλλά πιστεύω ότι έχει νόημα στον τομέα αυτό να προταθεί μια ευρωπαϊκή οδηγία. Και αυτό γιατί πιστεύω ότι οι διάφοροι πάροχοι δεδομένων, διαστημικών δεδομένων και δορυφορικών δεδομένων χρειάζονται ένα κοινό πλαίσιο προκειμένου να μπορέσουν να τοποθετηθούν σωστά και σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό με τα τρίτα κράτη. Αυτό φυσικά δεν επιτρέπεται να προκαλέσει πιο πολύ γραφειοκρατία. Όποιο ανησυχεί για το ότι θα αναγκαστούν και 28 χώρες ε, να δημιουργήσουν μια εθνική υπηρεσία ανεξάρτητα από το αν δραστηριοποιούνται στον τομέα των διαστημικών και δορυφορικών δεδομένων, πρέπει να ησυχάσει. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Όποιος έχει και κάνει αγοραπολισίες και συναλλαγές τέτοιες, ε, θα πρέπει να δημιουργήσει μια τέτοια υπηρεσία. Αυτό είναι λογικό. Αλλά θέλουμε να κάνουμε και κάποιες βελτιώσεις στην οδηγία. Αυτό θα είναι, αυτή θα είναι η δουλειά μου τις επόμενες εβδομάδες. Προσβλέπω σε αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις παρατηρήσεις σας και ελπίζω και είμαι σίγουρη άλλωστε ότι θα είναι και πολύ καλή η δουλειά από πλευρά του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα, να σας αναφέρω ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών, συγγνώμη, ανταλλαγή απόψεων 15 και 16 Ιουνίου. 15, 16 June. okay. 15 και 16 Ιουνίου. Εξέταση του σχεδίου έκθεσης. 17 Ιουνίου κατά πάσα πιθανότητα η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών, άρα να είμαστε έτοιμοι. Δεν θα έχουμε πολύ χρόνο μεταξύ της εξέτασης και της κατάθεσης, της προθεσμίας κατάθεσης τροπολογιών. Να παρακολουθούμε λοιπόν το θέμα, να παρακολουθούμε τις συνεδριάσεις των σκιωδών. Κυρία εισηγήτρια, έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας ακόμα τρεις μήνες να το συζητήσουμε το θέμα αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ασφαλώς. Και ασφαλώς και επηρεάζει και την ψηφιακή ατζέντα, την ενεργειακή ένωση, τα ευφύη δίκτυα και πάρα πολλά ζητήματα. Όπως είπατε και εσείς κυρία εισηγήτρια. Πολύ σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Και τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ευκαιρίες πράσινη ανάπτυξη για τι μικρόμεσες επιχειρήσεις. Είναι το 6. Αλλά ο Φίλιπ Ντεμπάκερ, ο εισηγητή μας, θα καταφτάσει σε λίγα λεπτάκια. Δεν είναι ακόμα εδώ. Άρα θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγο. Τρία λεπτάκια. Πέντε. to is slightly too long, but okay, we can stay even Πέντε λεπτά να περιμένουμε. Σημαντικό θέμα. Ευκαιρίες πράσινης ανάπτυξης. Short break. Okay, it's very, very. Dear colleagues, ladies and gentlemen, our colleague uh, Philip, Philip de Backer is Ο Φίλιπ Ντεμπάκερ είναι πολύ πιο γρήγορος και αποτελεσματικός από ό,τι νομίζαμε, γιατί ούτε καν πέντε λεπτά δεν χρειάστηκε να λείψει. Δύο λεπτά λοιπόν έλειψε. Και περνάμε λοιπόν στο θέμα της ευκαιρίας πράσινης ανάπτυξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ συνάδελφοι. 183 τροπολογίες έχουν κατατεθεί για την έκθεση αυτή. Η πρώτη άλλωστε της θητείας για τις μικρομεσαίες και την πράσινη ανάπτυξη. Πρότεινατε και κάποιες ε, συμβαστικές τροπολογίες με τους κοιόδης. με μεγάλη ανυπομονησία περιμένουμε να ακούσουμε τι έχει να μας πείτε. Είναι η πρώτη συζήτηση για το θέμα αυτό στην ε, Επιτροπή μας. Πείτε μας λοιπόν τι έγινε. Ο συνάδελφος κύριος Ντεμπάκερ έχετε το λόγο για να μας παρουσιάσετε τις τροπολογίες και τις συμβαστικές τροπολογίες. Uh, σας ευχαριστώ πάρα πολύ πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Χαίρομαι που μπορώ να σε ενημερώσω για την πρόοδο που έχει σημειωθεί όχι μόνο από τους συναδέλφους μου που κατέθεσαν τροπολογίε στο σχέδιο της έκθεσής μου το οποίο παρουσίασα πριν από κάποιες εβδομάδες στην Επιτροπή μας αλλά θα σας ενημερώσω και για τις απόψεις άλλων συναδέλφων. Είχαμε μάλιστα και μία πρώτη συνάντηση για αυτές τις τροπολογίε για να ε, τύχουμε 180 τροπολογίες κατατέθηκαν και πρέπει να πω ε, πολλές από αυτές αποτελούν βελτίωση του σχεδίου έκθεσης. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτές αποτελούν υπεραξία και τις δεχτήκαμε τις περισσότερες από αυτές ε, και προσπαθήσαμε να επιτύχουμε συμβαστικές στην Την Πέμπτη είχαμε την πρώτη συνεδρίαση των σκιωδών και κανονικά ε, τις πρώτες συμβαστικές θα τις ολοκληρώσουμε τις επόμενες ημέρες. Νομίζω λοιπόν σε γενικές γραμμές ότι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε μια καλή συμβαστική πρόταση. Θα αναφέρω πολύ σύντομα ορισμένα βασικά θέματα των τροπολογιών ε, και κάποιους συμβιβασμού που επιτύχαμε. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, ε, χάρηκα πάρα πολύ που είδα ότι η μεγάλη πλειοψηφία των μελών συμμερίζονται τη δική μου την άποψη για το σχέδιο της έκθεσης και τη δομή του. Και αυτό βοήθησε για να εστιάσουμε την προσοχή μας σε κάποια θέματα που εκκρεμούν. Προσπάθησα λοιπόν να διατηρήσω την ίδια δομή του εγγράφου για λόγους σαφήνειας. Ε, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή δομή αυτή της έκθεσης. Επιλέξαμε να μην απομακρυνθούμε από διάφορα θέματα ε, που έχουν σχέση με προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αγορά και εστιάσαμε την προσοχή μας στο τι μπορεί να επιτευχθεί στην πράσινη οικονομία. Για μένα λοιπόν η έκθεση είναι η αναζήτηση δυνατοτήτων για να καλυφθεί το χάσμα και ε, για να αναπτυχθεί πλήρως η πράσινη ανάπτυξη. Επίσης επιτύχαμε συμβαστική πρόταση όσον αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Το θέμα εξακολουθεί να είναι επίκαιρο ε, όχι μόνο για τις μικρομεσαίες αλλά και για άλλες επιχειρήσεις και έτσι ε, προσπαθήσαμε να εστιάσουμε την προσοχή μας στο τι μπορεί να γίνει κυρίως ε, για την κατάθεση νέων προτάσεων. Ε, προσπαθήσαμε να διευκρινίσουμε τι μπορεί να γίνει στον κύκλο ζωής αυτών των επιχειρήσεων, κυρίως όταν φτάνουν στη χρηματοδότηση. Προσπαθήσαμε επίσης να δώσουμε και κάποιες προτάσεις για ευρύτερες δυνατότητες χρηματοδότησης. Το τρίτο επί το οποίο εστιάσαμε έχει σχέση με όλα αυτά, είναι λίγο ευρύτερο είναι μια πρωτοβουλία που προέκυψε όχι μόνο μετά από συζητήσεις με συναντέλφους αλλά και με άμεσα εμπλεκόμενους. Το βασικό θέμα είναι ε, πώς θα αντιμετωπιστούμε τη διαχείριση της γνώσης ε, ε, και επίσης και πολλά άλλα στοιχεία τα οποία έχουν σχέση με την εικόνα που προέκυψε όταν αρχίσαμε να συζητάμε. Το τελευταίο θέμα βέβαια ήταν ότι όλα αυτά έχουν άμεση σχέση με την πράσινη οικονομία. Γνωρίζουμε ότι οι Επίτροποι έχουν κλείσει τη, τη δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία. Μας είπαν ότι θα καταθέσουν νέα δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία, για την πράσινη ανάπτυξη. Ε, αυτά όλα θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο και στις μελλοντικέ συζητήσεις. Όλες αυτές λοιπόν οι διαφορετικές πρωτοβουλίες βοηθούν στο να κατανοήσουμε καλύτερα τις νέες τεχνολογίες και επίσης βοηθούν και στην ανακούφιση από το διοικητικό άχθος. Προέκυψε ε, σαφής πλειοψηφία στις συζητήσεις και όλα αυτά βέβαια πρέπει να συνδυαστούν. Ανακεφαλαιώνοντας, οι τροπολογίες που πήραμε ήταν πολύ χρήσιμες, ε, κατέστησαν τις, ε, την έκθεση πολύ καλύτερη και είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσουμε επίσης να υποβάλουμε μια πολύ καλή έκθεση που θα είναι ένα σημαντικό μήνυμα όχι μόνο ανάμεσα και ε, στους ίδιους τους θεσμούς αλλά και γενικότερα στην αγορά. Προσβλέπω και σε καλύτερη συνεργασία ε, τις επόμενες μέρες για να ολοκληρώσουμε την έκθεση. Πολύ ωραία λέει ο Πρόεδρος. Τώρα, οι σκιώδεις συζητητές παρακαλώ. Ε, θα ήθελα και εγώ, λέει ο κύριος Ρουιμπίχ, να ευχαριστώ καταρχήν θερμά τον εισηγητή, γιατί το κλίμα των συζητήσεων είναι πολύ επικοδομητικό και νομίζω στο κοινοβούλιο μας αυτή είναι η απόλυτη προϋπόθεση για να επιτύχουμε καλά αποτελέσματα. Η έκθεση φέρει τον τίτλο «Δυνατότητες ανάπτυξης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως στον τομέα της αηφορίας». Όσον αφορά την ανάπτυξη, αυτό που παίζει ρόλο είναι να προσφέρονται κίνητρα. Τι είδου κίνητρα μπορούμε να ε, προσφέρουμε και ενώ η Επιτροπή Περιβάλλοντος κατά κανόνα δουλεύει με κυρώσεις, εμείς θέλουμε να βρούμε τα κίνητρα γιατί ε, αυτά είναι πολύ πιο σημαντικά. Οι κυρώσεις δεν προσφέρουν ανάπτυξη, αλλά οδηγούν στην ανεργία. Γι' αυτό λοιπόν για μας είναι σημαντικό ε, στα κράτη-μέλη οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μεριμνούν έτσι ώστε οι επιπτώσεις της ε, ευρωπαϊκής ε, νομοθεσίας να ελέγχονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί κανείς να δει κατά πόσον η ανάπτυξη ε, στις εξαγωγές, κατά πόσον η ανάπτυξη ε, θα οδηγήσει σε μεγαλύτερο κεφάλαιο κινδύνου στις επιχειρήσεις γιατί βεβαίως θα καταβληθούν ε, περισσότερες προσπάθειες εξαγωγών άρα δηλαδή και μεγαλύτερος κίνδυνος ε, και κατόπιν τούτου θα πρέπει να υπάρχει στις επιχειρήσεις κεφάλαιο κινδύνου έτσι ώστε να διασφαλίζεται και η χρηματοδότηση στις εξαγωγές αλλά και στις καινοτομίες. Θεωρώ ότι αυτή είναι η βασική έννοια. Έχουμε πάρει πάρα πολλές και καλές ε, ε, θετικές τροπολογίες πραγματικά εξεπλάγινε για το πόσο πολλές και καλές προτάσεις κατατέθηκαν και σε κάποιες όπου δεν είμαστε ακόμα, τα, ακόμα σίγουροι θα δούμε ε, πώς μπορούμε να καταλήξουμε κάπου με τον εισηγητή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Κόφορτ εκ μέρους των Σοσιαλδημοκρατών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, θα ξεκινήσω και εγώ ευχαριστώντας τον εισηγητή για την πάρα πολύ καλή του έκθεση και συνεργασία, πολύ καλή και δουλειά με τις ε, τροπολογίες. Όλα αυτά έχουν σχέση βεβαίως με τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με την πράσινη οικονομία. Νομίζω ότι η υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι καθοριστική σημασίας. Βεβαίως ε, μέσα στην έκθεση πάρα πολλά ε, είχαν σχέση με την πρόσβαση στο κεφάλαιο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και επίσης χαίρομαι που εξετάζει τώρα και ο πράσινος τομέας στο σύνολό του. Νομίζω λοιπόν ότι οι τροπολογίες και οι συμβαστικές προτάσεις ενισχύουν την έκθεση. Χαίρομαι λοιπόν για το πλαίσιο αλλά και για το πώς οι τροπολογίες μπορούν να ενταχθούν στην πράσινη οικονομία. Κατόπιν υπάρχουν κάποια θέματα που έχουν απομείνει, αλλά θα επιληθούν. Για μένα, ας πούμε, είναι σημαντικό ότι αν υπάρχει δημόσιο ενδιαφέρον για την υποστήριξη μη όριμων τεχνολογιών, αυτό το συζητήσαμε και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε κάποια συμβαστική λύση επ' αυτού. Δεν θέλω να μακρηγορήσω πρόεδρε γιατί νομίζω ότι καταλήξαμε σε μια πολύ καλή πρόταση. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους και εισηγητές. Ξέρω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα γιατί μερικοί από εμά δεν ήμασταν εδώ την προηγούμενη εβδομάδα αλλά κατορθώσαμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευκαιρίε πράσινη ανάπτυξη για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Κανεί άλλο θέλει να πάρει το λόγο, δεν βλέπω. Από Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποιον έχουμε. Ποιος εκπροσωπεί την Επιτροπή. Our rapporteur, dear colleague, dear colleague. Ο εισηγητής μας. Αγαπητέ συνάδελφε Τεμπάκερ, παρακαλώ μπορείτε να δευτερολογήσετε και να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση αφού τοποθετήθηκαν οι σκιώδεις Πάρα πολύ καλό ότι δεν έχουμε θέματα εδώ επίμαχα και θα έχουμε και τις τροπολογίες, οπότε όλοι μαζί ε, θα βγάλουμε συνεργασία. όποιος ήθελε να έχει αντιρρήσει, σα το είχε πει μέχρι τώρα. Πέραν των αστείων πάντω, ευχαριστώ για το όσα είπατε. Έχουμε ακόμα ένα-δύο σημεία τα οποία θα πρέπει κάπως να τα ξεσκονίσουμε, αλλά τέλος πάντων. Θα πρέπει να δούμε με την χρηματοδότηση πώς όλα αυτά θα μπορούν να ενσωματωθούν στην πράσινη οικονομία περισσότερο από ό,τι πριν. Και αυτό το οποίο εκκρεμεί το ανέφερε ο σοσιαλιστής συνάλφος στον αφορά τις ε, ανώνυμες τεχνολογίες. Βεβαίω και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η προβληματική, αλλά τελικά νομίζω ότι όλοι στο ίδιο κατατείνουμε. Δηλαδή πώς, τι θα γίνει με τις ε, προμήθειες, να δώσουμε ευκαιρίες σε νέες τεχνολογίες, αλλά να μην παρισφρήσουν και να μην επιδοτηθούν από τα κράτη-μέλη ε, κάποιες ανώριμες τεχνολογίες. Πάντως έχουμε περικοπές ε, λόγω της λιτότητας και νομίζω ότι απλώς είναι το θέμα του να βρούμε μια διατύπωση που να αντικατοπτρίζει ότι όλοι θέλουμε το ίδιο και νομίζω ότι τις επόμενες ώρες, τις επόμενες μέρες θα σας στείλω κάποια συνδυαστικά κείμενα και θα δείτε ότι ε, ή επιλήθηκαν τα θέματα τα οποία είναι πιο επίμαχα ή θα έχω βρει μια καινούργια διατύπωση που και εδώ και στην Ολομέλεια τελικά τους βρουν όλους σύμφωνους γιατί όλοι συμφωνούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική σημεία για την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Επίσης, συνέχεια όσων είπε στην αλήθεια, πρέπει να πούμε ότι οπωσδήποτε και υπάρχει πρόθεση υποστήριξης των ΜΜΕ ε, γενικώ και κατά συγκεκριμένο τρόπο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι ευκαιρία δημιουργήσει θέσεων απασχόληση για του ε, συμπολίτε μα. Γι' αυτό και θέλουμε την πράσινη ανάπτυξη. Uh, η ψήφιση του σχεδιοκειμένου θα γίνει στις 14 Τετάρτου. Στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής μας. Αύριο, η ώρα, θα συνεδριάσουν οι συντονιστές. Αλλά η Επιτροπή, όλοι μας δηλαδή, θα αρχίσει να συνδέεται στις 10 η ώρα και θα έχουμε τις ψηφοφορίες. Φέρτε τις ε, κάρτες τελευταίες ψηφοφορίας. Σας ευχαριστώ, τα πούμε αύριο.